Hello, nice to see you. Hello. Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μόλις ήρθα από την Επιτροπή των Περιφερειών και τα μέλη της ε, ενδιαφέρονται πάρα πολύ για τη δέσμη μέτρων για την ενέργεια, καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους έχουν πολλά ερωτήματα για τις ευθύνες πόλεις, για όλα αυτά τα θέματα. Είναι λοιπόν η σημερινή ακρόαση πολύ ενδιαφέρουσα και για μας και για την Επιτροπή των Περιφερειών. Ας αρχίσουμε όμως τη δημόσια ακρόαση με θέμα καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους. Θα χωριστεί σε δύο κομμάτια το ο σχεδιασμός της αγοράς ενέργειας για το μέλλον και ποιες αλλαγές είναι αναγκαίες και το δεύτερο τμήμα είναι η συμπερίληψη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην αγορά, ποιες είναι ευκαιρίες, ποια είναι τα εμπόδια. Η ακρόαση φυσικά είναι Αποτέλεσμα της δημοσίευσης 30 Νοεμβρίου του 2016 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 8 νομοθετικών προτάσεων, το μεγαλύτερο νομοθετικό πακέτο που έχει δημοσιεύσει μέχρι τώρα. Κάποιες, αφορούν, κάποιες προτάσεις αφορούν την ενεργειακή απόδοση, τις ανανεώσιμες, σε γενικές γραμμές δηλαδή. Ε, θέματα ενεργειακής διακυβέρνησης και νέου σχεδιασμού της αγοράς ενέργειας. οι οχτώ νομοθετικές προτάσεις χωρίζονται σε δύο κύριους τομείς. Ο κάθε ένας θεωρείται μια δέσμη μέτρων, όχι λοιπόν και οι οχτώ μαζί, αλλά τέσσερα και τέσσερα. Το πρώτο κομμάτι αναμένουμε να το έχουμε ολοκληρώσει τον Οκτώβριο και το δεύτερο τον Νοέμβριο. Προσπαθούμε λοιπόν μέχρι τότε να ενημερωθούμε όσο το δυνατόν πληρέστερα Γι' αυτό η δημόσια αυτή ακρόαση νομίζω πως είναι πολύ επίκαιρη. Καλωσορίζω λοιπόν όλους τους προσκεκλημένους μας από το πρώτο και το δεύτερο πάνελ. Χαίρομαστε πολύ που ήρθατε. Ε, και περνάμε τώρα στο πρώτο πάνελ, ο σχεδιασμός της αγοράς ενέργειας για το μέλλον. Ποιες αλλαγές χρειάζονται. Η αγορά ενέργειας χρειάζεται αλλαγές τόσο στον τομέα του φυσικού αερίου όσο του ηλεκτρισμού και αυτή η δέσμη μέτρων αφορά κυρίως τον ηλεκτρισμό. Ας μην ξεχνάμε όμως και το φυσικό αέριο, το οποίο ε, έχει ένα μεγάλο μερίδιο της αγοράς. Χρειάζεται, είναι, είναι αναγκαία η συμβατότητα ανάμεσα στις δύο αυτές πηγές ενέργειας. Είναι πολύ σημαντικό επίσης και για την ε, λειτουργία της ενίας αγοράς για τις εκπομπές αερίων, για παράδειγμα. Υπάρχουν άλλες ε, ανώτατες τιμές για το φυσικό αέριο και άλλες για ε, τον ε, ηλεκτρισμό. Εδώ θα επικεντρωθούμε λοιπόν στον ηλεκτρισμό, χωρίς να ξεχνάμε και το φυσικό αέριο. Πρώτος προσκεκλημένος, ο κύριος Τομπίας Παόλουν, είναι επικεφαλής στρατηγικής από την European Energy Exchange. Μία από τις ηγετικές πλατφόρμες ενέργειας αυτή τη στιγμή και η EEX επίσης ασχολείται με εμπορία ρήπων. Όχι μόνο δηλαδή με ηλεκτρισμό, με ενέργεια, αλλά και με εμπορία εκπομπών. Είναι λοιπόν πολύ σημαντική η αγορά αυτή και η πρόταση σχετικά με το σύστημα εμπορία εκπομπών συνδέεται άμεσα με αυτή. Θα ήθελα λοιπόν να σας δώσω το λόγο και να σας ε, παρακαλέσω να μην υπερβείτε τα 7 λεπτά, διότι μετά τις ε, παρουσιάσεις σας θα έχουμε και συζήτηση. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αγαπητά μέλη της Επιτροπής, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να σας παρουσιάσω την άποψη του EEX για ε, τη δέσμη μέτρων σήμερα. Η δέσμη αυτή συμπεριλαμβάνει το ε, την πλατφόρμα ανταλλαγής ενέργειας βραχυ, ε, βραχυπρόθεσμης. Κοιτάζουμε έξι χρόνια μετά Πέρσι είχαμε συνολική ε, απόδοση 4.000 τεραβατορών. Καταφέραμε πολλά τα τελευταία χρόνια στην αγορά ενέργειας, χρειάζονται όμως να γίνουν περισσότερα, να αυξήσουμε την ορατότητα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τη συμμετοχή τους στην ε, αγορά ενέργειας, αλλά και να βελτιώσουμε την ήδη καλή λειτουργία της αγοράς τώρα. Το το πακέτο αυτό, η δέσμη μέτρων, ε, νομίζω πως είναι καλό να, να το δούμε λίγο πιο γενικότερα. Λίγο μετά την ε, ψηφοφορία, το δημοψήφισμα για τον Brexit, ε, δημοσιεύθηκε αυτή η δέσμη μέτρων και πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση της συνέχειας, το τι θα κάνουμε μετά στο χώρο της ενέργειας. Γι' αυτό λοιπόν η δέσμη μέτρων νομίζω πως είναι μια ευκαιρία να αλλάξουμε όραμα, να αλλάξουμε τους στόχους και να δούμε πώς μπορούμε να εποφεληθούμε όλοι από την ε, συγκέντρωση όλων των πηγών ενέργειας σε μία αγορά, έτσι ώστε να επωφεληθούν οι πολίτες και η κοινωνία γενικότερα. Η δέσμη μέτρων έχει δώσει κάποιες απαντήσεις, αλλά σε ορισμένους τομείς νομίζω πως χανόμαστε στις λεπτομέρειες. Γι' αυτό είναι καλό το όραμα να είναι σαφές, ξεκάθαρο, οι ευθύνες που θα ε, δοθούν να είναι και επίσης ε, σαφής έτσι ώστε το όραμα να, για το μέλλον να είναι και αυτό σαφέστερο. Η αγορά ενέργειας χωρίζεται σε τρεις πυλώνες. Καταρχάς συντονισμός που καθορίζεται από τις τιμές της αγοράς, από τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας, από τις επενδύσεις. Μετά υπάρχουν μεγάλες και ρευστές ζώνες, κατηγορίες τιμών και γι' αυτό χρειάζεται ε, να χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και ανταγωνιστικότητα. Μετά, οι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια πρέπει να ενσωματωθούν πλήρω στην αγορά ενέργεια, έτσι ώστε να αποφύγουμε ε, στρεβλώσει τη αγορά, των τιμών κτλ. Αυτό είναι το δικό μα όραμα μακροπρόθεσμα για την ε, αγορά ενέργεια. Μέχρι τώρα έχουν γίνει αρκετά και όπως σας είπα είναι ανταγωνιστική αγορά ενέργειας. Η γερμανική και αυστριακή ζώνη τιμών είναι αυτή τη στιγμή η πιο δυνατή στην Ευρώπη, πιο ανταγωνιστική, όμως αναδύονται και άλλες αγορές, ε, πολλά υποσχόμενες. Το όραμα λοιπόν από την δέσμη μέτρων μπορεί να χτιστεί πάνω σε αυτά που ήδη έχουμε διαθέσιμα σήμερα. Τώρα υπάρχουν τέσσερις τομείς που εντοπίσαμε και θα ήθελα να σας τους παρουσιάσω και να ακούσω επίσης και το πώς εσείς το, τους εκτιμάτε. Καταρχάς, οι τιμές από την ίδια την αγορά, όπως ε, σας είπα, αναφέρονται σε αυτό το πακέτο, είναι ορατές, χρειάζεται να είναι καθαρές και, ευ, και ευδιάκριτες οι τιμές έτσι ώστε να αποφύγουμε στρεβλώσεις της ε, αγοράς. Να τονίσω όμως ότι ο ορισμός των ανώτατων, ορίων, ε, ανώτατων τεχνικών ορίων είναι καλύτερο να είναι αρμοδιότητα των ε, χρηματιστηρίων ενέργειας, των αγορών ενέργειας και των ε, φορέων εκεί. Μετά, αντισταθμιστικές δυνατότητες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο του, ε, της δέσμης μέτρων ε, για το χειμώνα. Εδώ υπάρχει λιγότερη ανταγωνιστικότητα, λιγότερη διαφάνεια. Και μάλιστα στην αγορά ενέργειας, στο χρηματιστήριο ενέργειας υπάρχουν νέα ε, συστήματα, νέα εργαλεία που είναι αφιερωμένα στις ανανεώσιμες και μπορούν να βοηθήσουν στην περαιτέρω προώθησή τους. Μετά, ο επόμενος τομέας μας ανησυχεί αρκετά. Είναι δηλαδή το πώς θα οριστούν οι ζώνες, ε, προσφορών. Σε σχέση με τα προηγούμενα νομοθετικά πακέτα, παρατηρήσαμε ορισμένες ανισορροπίες, ε, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με αυτές τις ζώνες υποβολής προσφορών. Στην ουσία, εδώ έχουμε μια διαφορετική οπτική γωνία. Προτείνεται ένα άλλο μοντέλο, αλλά η, αγορά, η χονδρική αγορά ενέργειας πρέπει να είναι ανταγωνιστική και διάφανη στο δυνατόν περισσότερο. Τέταρτος τομέας έχει να κάνει με τους ε, μηχανισμούς χορτικότητας ε, ενέργειας. Εδώ φυσικά πρέπει να γίνονται σεβαστές οι εθνικές ε, αρχές, η εθνική νομοθεσία και πρέπει να υπάρχουν και εδώ σαφείς ορισμοί Πρέπει όμως να τονίσουμε ότι η αγορά ε, ικανοτήτων ηλεκτροπαραγωγικής ενέργειας πρέπει να είναι ανοιχτή και για διασυνοριακούς ε, παράγοντες. Έκτος τομέας, πέμπτος με συγχωρείτε, είναι η συμπερίληψη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην αγορά ενέργειας. Και εδώ το κύριο σκεπτικό είναι ότι οι τιμές δεν πρέπει να στρεβλώνουν τα σήματα που μας δίνει η αγορά, γι' αυτό, χρειάζονται γι αυτό χρειάζεται οριοθέτηση. Εδώ είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος των ε, χρηματιστηρίων, των ε, short-term αγορών. Μετά, συντονισμός. Ο συντονισμός ανάμεσα στις περιφέρειες, ανάμεσα στους διάφορους τομείς πολιτικής. Η περιφερειακή συνεργασία είναι πάρα πολύ σημαντική έτσι ώστε να αναπτυχθεί μια ανταγωνιστική, ολοκληρωμένη ε, ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, συμπεριλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις εδώ. Γι' αυτό ε, στο πακέτο αυτό τη δέσμετρο για το χειμώνα είναι πολύ σημαντική αυτή η συνεργασία. Υπάρχουν κάποια περιφερειακά κέντρα τα οποία ε, σε ό,τι αφορά την επιχειρησιακή τους ε, λειτουργία έχουν κάποια προβλήματα. Μετά θα ήθελα να τελειώσω λέγοντας ότι πρέπει να γίνει σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στο, ε, στην ενεργειακή δέσμη μέτρων και στο, στη δέσμη του για το κλίμα. Αυτά τα 50 γραμμάρια ανά κιλοβατόρα, ο κανόνας αυτός τα 550, με συγχωρείτε, είναι ε, κάτι που δεν συμφωνεί με το άλλο. Πρέπει να υπάρχει ένας κοινό στόχος, μια κοινή τιμολόγηση, ε, κοινό όρεμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Να δώσουμε τώρα το λόγο στην κυρία Νίσ από τον Ένσο Ι. Να πάρει το λόγο. Σας επενθυμίζω ότι ο Ένσο Ι δημιουργήθηκε βάσει της τρίτης ε, νομοθετικής ε, δέσμης το 2009. Και εκπροσωπείται τώρα 42 TSOs από 35 χώρες σε όλη την Ευρώπη. Επομένω, ε, δεν αφορά αυτό μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορείτε να δώσετε μια ευρύτερη εικόνα για τον σχεδιασμό της αγοράς από πλευράς ε, παρόχων που από ό,τι φαίνεται εκεί έγκυται στο μεγαλύτερο βαθμό η εστρική μας ε, αγορά ενέργειας, γιατί είστε έντσο ε, όχι έντσο G, αλλά και πάλι δεν βρίσκεται αυτό σε αντιδιαστολή. Έχετε πολύ καλές σχέσεις. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω εγώ να μιλήσω πιο γρήγορα για να μην χαθεί χρόνο. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίε και κύριοι, σα ευχαριστώ πολύ ε, που με καλέσατε εδώ και εμένα και τον οργανισμό μου για αυτή τη σημαντική συζήτηση. Όπω είπε ο κύριος Μπούζακ, υπάρχει μόνο μία αγορά ενέργειας και ακόμα και αν έχουμε τον ENSO E και τον ENSO G, είναι σαφές ότι το θέμα, το μέλλον μάλλον θα είναι η σύζευξη, σύνδεση κλάδων και στην Ευρώπη θα έχουμε εξαιρετικές, έχουμε εξαιρετικές υποδομές και στην ηλεκτρική ενέργεια και στο φυσικό αέριο. Πρέπει να τα πλουταστοποιήσουμε σε ό,τι αφορά τους πόρους. Για την ηλεκτρική ενέργεια, όπως είπε ο κ. Μπούσεκ, εμείς υπερβαίνουμε τα ευρωπαϊκά ε, σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 42 μέλη, πολύ σημαντικά τα μέλη μας. Η ευρωπαϊκή διασυνοριακή διάσταση της ηλεκτρικής ενέργειας μας αναγκάζει να το εξετάζουμε όλο αυτό ε, σε, από μια περιφερειακή προσέγγιση και διάσταση, μη εθελοντική, δεσμευτική, περιφερειακή και ευρωπαϊκή διάσταση. Σε ό,τι αφορά την μετάβαση, την ενεργική μετάβαση, η χειμερινή δέσμη ή, ε, όπως αποκαλείται τώρα πολύ ωραία, καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους, είναι μια δέσμη μέτρων που θέλει να διασφαλίσει βιώσιμη και ασφαλή και ανταγωνιστική ε, ενέργεια και ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο, σύνδεση με τον κλάδο των μεταφορών και τη φιλοδοξία 45% ε, του ενεργειακού μείγματος αποκαλείται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι το 2030. Ο τίτλος εδώ είναι ποιες είναι οι απαραίτητες αλλαγές. Μία από τις αλλαγές που χρειαζόμαστε είναι να διατηρήσουμε ορισμένες ε, ήδη υφιστάμενες ε, ε, διατάξεις στο φιλόδοξο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ναι, στον, στο πρότυπο του ενεργού καταναλωτή. Ναι, χρειαζόμαστε ε, και συγκεκριμένα κίνητρα τιμολογικά ε, σε περίπτωση ε, περιορισμένων πόρων. Να άρουμε τυχόν ε, όρια τιμών, να έχουμε πιο εύκολη μετάβαση από τον ένα πάροχο στον άλλον, ένα πλαίσιο ετοιμότητας κινδύνου και χρειαζόμαστε και μία αξιολόγηση σε ό,τι αφορά τους ευρωπαϊκούς πόρους και την επάρκειά τους για να δούμε τι μπορούμε να διορθώσουμε στο μέλλον. Και βέβαια χρειαζόμαστε και μια ιδιαίτερα φιλόδοξη περιφερειακή συνεργασία, προκειμένου να πετύχουμε τους στόχους μας μέχρι το 2030. Θα ήθελα να σταθώ στα περιφερειακά επιτεύγματα, καθώς υπήρξε μια μακρά συζήτηση για το, σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα το παράδειγμα της κεντρικής Ευρώπης. Η ολοκλήρωση των συστημάτων ειδικής ενέργειας έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Βλέπετε Nordbalk, Litpol, Estlink, Νέα κράτη-μέλη λοιπόν, τα οποία έχουν ενταχθεί στο ευρύτερο ευρωπαϊκό σύστημα. Και βλέπετε εδώ, από πλευράς αγοράς, έχουμε περάσει στην σύζευξη των αγορών της Ανατολικής Ευρώπης, ε, ε, βόρειο-ανατολικής, ε, ε, δυτικής και τώρα θέλουμε να βάλουμε στόχο την σύνδεση και της ε, ε κεντρικής και ανα, ανατολικής Ευρώπης μέσα στα επόμενα χρόνια. Δεν θέλουμε ε, να υπάρχει χάσμα στην αγορά ενέργειας στην Ευρώπη. Και αυτό μας δίνει νέες ευκαιρίες, χαμηλότερες τιμές, περισσότερος ανταγωνισμός, βελτίωση στην αλυσίδα ρεφοδιασμού και μεγαλύτερη ολοκλήρωση για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τώρα, η επιφυλάξη μας, ο προβληματισμός μας. Σε ό,τι αφορά τους ε, κώδικες δικτύων, ήταν μια πολύ δύσκολη ε, και φιλόδοξη ε, διαδικασία που αφορούσε τον Acer μεταξύ του e, τον, του ENSO-G, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών. Θέλουμε να συνεχιστεί στο μέλλον αυτή η προσπάθεια και βλέπουμε όμως ότι στη δέσμη δεν υπάρχει σχεδόν ούτε καν αναφορά, ενώ αποτελούν προτεραιότητα. Ε, θα πρέπει, παρότι υιοθετήθηκαν την περασμένη εβδομάδα, να υλοποιηθούν μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. Πρέπει λοιπόν να προετοιμαστούμε, να προετοιμάσουμε το έδαφο. Σε ό,τι αφορά τα περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα, στηρίζουμε απολύτω το να είμαστε φιλόδοξοι σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και σε ό,τι αφορά τη συνεργασία των τοπικών και περιφερειακών φορέων. Όμω, δεν δεχόμαστε μια δεσμευτική διαδικασία λήψη αποφάσεων σε τέτοιε νέε δομέ που δεν έχουν κάποιο αντιστάθμισμα σε εθνικό κράτος μέλος. Όπου δηλαδή δεν υπάρχει περιφερειακός, ε, περιφερειακή ρυθμιστική αρχή και αυτό δημιουργεί ε, μεγάλο πλεονέκτημα ίσως προς τα κράτη-μέλη. Σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό της αγοράς, έχουμε κάποιους προβληματισμούς που έχουμε ε, επισημάνει στην πρόσφατη έκθεσή μας. Και σε ό,τι αφορά την ολοκλήρωση της αγοράς χοντρικής και λιανικής, θεωρούμε ότι πρόκειται για σημαντικά βήματα, αλλά υπάρχει κίνδυνο στήριξη των τοπικών αγορών και αυτό μας απομακρύνει από την ολοκλήρωση της αγοράς χανδρικής και λιανικής. Συνοπτικά, αυτό σημαίνει ότι οι πελάτες, οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να ε, δραστηριοποιούνται σε όλη την ευρωπαϊκή αγορά και όχι μόνο στην τοπική τους αγορά. Θέλαμε λοιπόν να υπάρχει το δικαίωμα διασυνοριακής ανταλλαγής. Η νέα όμως ε, επικαιροποίηση, η νέα εκδοχή θέλει να πάρει αυτή την ευελιξία προς ε, ολόκληρη την αγορά. Ευχαριστώ. Madam, and now I would like to ask Mr. Ευχαριστώ. Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Μάτιας Μποκ, επικεφαλής της Αγόρα Energy Βέντε. Θα μας παρουσιάσει τις δικές του απόψεις. Ο κύριος Μποκ. Επί πάνω από δεκαέτη έχει συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήταν και στο επιτελείο του Γιάννη Ποτότσνικ, πρώην Επιτρόπου Περιβάλλοντος. αλλά και πιο παλιά, Επίτροπος ε, έρευνα και ανάπτυξη. Από αυτή την άποψη λοιπόν έχετε πολύτιμη πείρα στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος και του κλίματος. Έτσι, η θέση σας και ως εκπροσώπου του Energy Event που σημαίνει ότι υπάρχει μια μετάβαση, μεταβατική περίοδο για την ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά και ενδιαφέροντα για μα. Παρακαλώ. Ε, σας ευχαριστώ. Και σα ευχαριστώ για την πρόσκλησή σα να παρουσιάσουμε τι δικέ μα απόψει. δεδομένου ότι είμαστε μια δεξαμενή σκέψη που ε, δράζεται στο Βερολίνο, χρηματοδοτούμαστε από φιλανθρωπικά ιδρύματα, δεν έχουμε κανένα εμπορικό συμφέρον σε αυτή τη συζήτηση. Απλά μα έχουν αναθέσει οι ιδρυτέ μας να σκεφτόμαστε ε, για το μέλλον ξεκινώντας με την ε, γερμανική ενεργειακή μετάβαση που είναι ένα πολύ μακροπρόθεσμο project αλλά όλο ένα και περισσότερο ε, προβληματιζόμαστε για το, ε, το ευρωπαϊκό επίπεδο και τώρα ξεκινάμε συζητήσεις και με τις διεθνείς αγορές. Τώρα εγώ θα εστιάσω σε συγκεκριμένα θέματα κλειδιά που θεωρούμε ότι είναι σημαντικό σε αυτό το πολύ περίπλοκο χειμερινό πακέτο δέσμη μέτρων και θέλω να ξεκινήσω τονίζοντας ότι φυσικά ό,τι και αν συμβεί στην, ε, σε επίπεδο της Ένωσης, σε εθνικό επίπεδο όσον αφορά το την προστασία του κλίματος και την ενέργεια, η συνεργασία ε, φέρνει πολύ καλύτερα αποτελέσματα από τη μοναχική δράση. Πιστεύουμε λοιπόν ότι το πακέτο για την καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρώπους είναι μια σημαντική ευκαιρία ώστε να προχωρήσει η συζήτηση περί της Ευρώπης σε εθνικό επίπεδο με θετικό τρόπο και ώστε να τονίσουμε τι μπορεί να προσφέρει η Ευρώπη στους πολίτες της. Προχωρώ με τα εξή σημεία. Καλό είναι να πούμε ότι η Ευρώπη έχει ε, σημειώσει πολύ εντυπωσιακή πρόοδο προς μια εσωτερική αγορά ενέργειας. Τα επόμενα βήματα, όπως είπε και η προηγούμενη ομιλήτρια, είναι ο στόχος για την ανανεώσιμη ενέργεια που ορίστηκε από τους επικεφαλείς ε, κρατών ε, και κυβερνήσεων το 2014 σημαίνει 45% ανανεώσιμες μέχρι το 2030. Δηλαδή το ενεργειακό μείγμα πρέπει να είναι πολύ πιο ευέλικτο, σημαίνει αυτό τώρα μια βασική, μια βασικός άξονας της, της πρότασης της Κομισιόν είναι ακριβώς αυτή η μεγαλύτερη ευελιξία. Ενώ αν ταυτόχρονα δει κανείς το μείγμα, ενεργειακό μείγμα που ισχύει ήδη στην Ευρώπη, βλέπουμε ότι έχουμε υπερπαραγωγικότητα για την Ευρώπη, υπερπάρκεια για την Ευρώπη συνολικά και αν δούμε το μέλλον, ε, ε, και το πιο ευέλικτο μείγμα που χρειαζόμαστε για την Ευρώπη, πιθανότατα ορισμένες ε, δυνατότητες θα πρέπει να αποσυρθούν από το σύστημα και άρα να δημιουργήσουν έτσι χώρο για περισσότερη ευελιξία, πράγμα που θα επιτρέψει στις μεταρρυθμίσεις της αγοράς να είναι πιο αποδοτικές. Έχουμε τώρα κάποιες ενδιαφέρουσες ενδείξεις στις προτάσεις της Κομισιόν ότι επίσης θέλουν να εξετάσουν αυτό το θέμα της υπερπαραγωγικότητα στην πρόταση που ε, είναι πάνω-πάνω στο ιδέσμι. Η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι θα αρχίσει διάλογο με τα κράτη-μέλη που επιθυμούν να έχουν μια κοινωνικά δίκαιη μετάβαση σε, σε περιφέρειες ε, όπου υπάρχει εντατική χρήση άνθρακα και ε, εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Δεύτερο θέμα που θέλω να τονίσω είναι οι παρεμβάσεις στην ε, παραγωγή. Υπάρχουν σημαντικά κομμάτια της πρότασης Κομισιόν που αφορούν μηχανισμούς ε, παραγωγικότητας δυνατοτήτων και από τη δική μας προοπτική, όταν βλέπουμε δηλαδή την ευρωπαϊκή ενεργειακή μετάβαση, είναι πραγματικά κέριο αυτές οι παρεμβάσεις να είναι συνεπείς με την χαμηλότερη χρήση άνθρακα και τις ανάγκες ευελιξίας. Αυτό σημαίνει σύνδεση, απόδοση στην ενέργεια, τι συμβολή μπορούμε να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε τα θέματα της καταλληλότητας των πόρων και όλα αυτά θα πρέπει να είναι ένα απόσπαστο τμήμα των στρατηγικών για να αντιμετωπίσουμε τις ε, ανησυχίες περί καταλληλότητας των πόρων. Η πρόταση λοιπόν οθεί προς τη σωστή κατεύθυνση. Υπάρχουν σημαντικές ιδέες γιατί η καταλληλότητα των πόρων δεν σημαίνει μόνο ε, την ε, δυνατότητες αλλά και την πλευρά της ζήτησης. Πράγμα που μπορεί ωστόσο να ενισχυθεί στις διατάξεις για το πώς οι μηχανισμοί μηχανισμοί δυνατοτήτων θα σχεδιαστούν αν τα κρατημέλη θεωρήσουν ότι υπάρχει ζήτημα καταλληλότητας των πόρων. Σε αυτό το πλαίσιο επίσης πιστεύουμε, και αυτό είναι το πλαίσιο της προηγούμενης ομιλήτριας, ότι είναι καλή ιδέα να υπάρχει ένα πρότυπο απόδοσης εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα για να μπορούν να ελεγχθούν καλύτερα. Επόμενη μου παρατήρηση αφορά την ολοκλήρωση της αγοράς για τις όριμες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ε, φυσικά η ολοκλήρωση θα συνεχιστεί και από την πλευρά των κρατών η Κομισιόν πιέζει σκληρά ώστε να υπάρξει περισσότερη ολοκλήρωση. Έχουν υποχρεώσεις, έχουν ανταγωνιστικές, ε, ε, ανταγωνιστικούς ε, διαγωνισμούς στις κρατικές προμήθειες. Αν όμως θέλουμε να έχουμε 60 ευρώ ή περισσότερο από το ETS, δεν είναι ρεαλιστικό αυτό να θεωρήσουμε δηλαδή ότι θα έχουμε επενδύσεις που θα καθορίζονται από την αγορά στις ανανεώσιμες που πλήρως θα αποζημιώσουν ή θα αποσβέσουν τις επενδύσεις. Υπάρχουν αρκετές σχετικές μελέτες που το αποδεικνύουν αυτό. Αυτό σημαίνει ότι στις συζητήσεις για το σύστημα εμπορίας εκπομπών και το τι μπορούμε να αναμένουμε για από αυτό το σύστημα στη δεκαετία 2020-2030 Πιστεύουμε εντόνως, αν δούμε τα στοιχεία αυτά, ότι θα παραμείνει η σημασία ενός στεναρού πλαισίου για τις ανανεώσιμες. Αυτό σημαίνει ότι περιορίζεται ο κίνδυνο. και όταν περιορίζεται ο κίνδυνο, το κόστος για τον επενδυτή είναι όσο γίνεται πιο χαμηλό και φυσικά αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας εφόσον υπάρχουν ε, ανταγωνιστικές δυνατότητες για την ε, κατασκευή νέων ε, εγκαταστάσεων και τότε ε, μπορεί αυτό να επιβαρύνει την τελική τιμή του καταναλωτή και αυτό δεν είναι επιθυμητό. Γι' αυτό πρέπει να παραμείνει στεναρό το πλαίσιο ε, για τις ανανεώσιμες. Μια μου τελευταία μου παρατήρηση για το πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Ξέρω ότι είναι υποσυζήτηση από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το θέμα της μεταρρύθμισης του συστήματος εμπορίας εκπομπών. Το σχέδιο που βλέπετε εδώ, το γράφημα που βλέπετε, δείχνει ότι εκτός αν γίνουν ε, θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις ε, του ETS, ε, δεν μπορούμε να αναμένουμε στη δεκαετία 2020 με 2030 σημαντικές επενδύσεις. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Συζητάμε στο Κοινοβούλιο εδώ και πολύ καιρό για το σύστημα εμπορίας εκπομπών, πώς πρέπει να μεταρρυθμιστεί. Τώρα όμως θα ήθελα να δώσω το λόγο σε εσά, αγαπητά μέλη τη Επιτροπής, τους εισηγητές και σε όσους ζήτησαν το λόγο. Κυρίω ε, τους ε, εισηγητές. Αρχίζουμε με τον κύριο Κάριν, Σχεδιασμός της νέας αγοράς ενέργεια. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, πολύ ενδιαφέροντα αυτά που άκουσα. Έχω καταρχάς ένα σχόλιο και μια ερώτηση. Ε, να πω ότι άκουσα τον τελευταίο μιλητή και μου φάνηκε περίεργο που ακούω συνέχεια για τον κίνδυνο που έχουμε να μειωθεί ε, το κόστος. Αυτό όμως συνδέεται με την, με την μέγιστη χωρητικότητα. Όταν αυξάνεται η μέγιστη χωρητικότητα, μειώνεται και το κόστο. Γι' αυτό δεν καταλαβαίνω ακριβώ πώ το εννοείτε. Για όλου τώρα, εσά έχω μία ερώτηση. Ε, γνωρίζουμε ότι όσο οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας γίνονται πιο γνωστές, αυξάνονται, η χρήση, όσο αυξάνεται λοιπόν η χρήση τους, χρειάζεται όλο ένα και περισσότερο να υπάρχει ένα εφεδρικό σύστημα για όταν δεν θα υπάρχει αέρας, δεν θα υπάρχει ήλιος κτλ. Τώρα, μέχρι στιγμής Πώ το χειριζόμασταν αυτό. Ε, πληρώναμε κάποιον απλά για να είναι ε, έτοιμο αν τον χρειαστούμε να παρέμβει. Εγώ θέλω να ρωτήσω όμω το εξή Μπορεί η αγορά να παρέχει αυτό το εφεδρικό σύστημα, αυτή την εφεδρική ενέργεια έτσι ώστε να διασφαλιστεί ε, η συνέχεια της ηλεκτροδότηση, τη ενέργεια. Μπορούμε να περιμένουμε ας πούμε μία μέρα για να πάρουμε την εφημερίδα μα, αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε 20 λεπτά μέχρι να ξανανάψουν τα φώτα. Ε, αλλά πώ θα γίνει, πώ θα το κάνουμε αυτό με έναν καλύτερο τρόπο ε, από το να πληρώνουμε κάποιον απλά για να μην κάνει τίποτα σε περίπτωση που. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ όλου του προσκεκλημένους για τι εισηγήσεις του. Πρόκειται για ένα τεράστιο, μια τεράστια δέσμη μέτρων που θα εξετάσουμε και αν θέλουμε να τηρήσουμε τους στόχους που συμφωνήσαμε στο Παρίσι, δηλαδή θα πρέπει να φτάσουμε στην πλήρη πάυση της χρήσης του άνθρακα μέχρι το 2050 και πρέπει όλα ό,τι θα κάνουμε ε, να προχωρά προς αυτήν, την, αυτόν τον στόχο. Οι ενεργειακές αγορές πρέπει να αντιμετωπίσουν σημαντικές αλλαγές, πρέπει να ενσωματώσουν ανανεώσιμες ε, αποκεντρωμένες πηγές ενέργειας με διαφοροποιημένες και με χαμηλό κόστος ε, για τον καταναλωτή. Έχουμε και νέους φορείς, γι' αυτό και η αναθεώρηση αυτή είναι πολύ απαραίτητη. Γι' αυτό θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Πάολον ε, δύο ερωτήσεις όσον αφορά τις εγγύησεις προέλευσης. Ε, καταρχάς, ε, τη γνώμη του για το κατά πόσο η νέα νομοθεσία θα καλύψει τις αμφιβολίες για την προέλευση, για τη χρησιμοποιώ, αναφέρομαι στο συγκεκριμένο ε, ξέπλυμα, το πράσινο ξέπλυμα της ενέργειας, όπως το λέμε στην χώρα μου, και έπειτα για τις ενέργειες, τις ανανεώσιμες μπορούμε να έχουμε και εγγύησεις προέλευσης και τη, στην εκπρόσωπο τη ΕΝΤΣΟ θέλω να τη ρωτήσω για τις προκλήσεις των διασυνδέσεων, κυρίως σε χώρε όπω η Ισπανία, ώστε να έχουμε περισσότερες δυνατότητες για τι ανανεώσιμε. Επίσης θα ήθελα να γνωρίζω ποιο έχει την ίστατη ευθύνη ε, για το συντονισμό ανάμεσα στους ε, TSO σε περιφερειακό επίπεδο. Σα ευχαριστώ πολύ. Adam Σας ευχαριστώ πολύ. Μία ερώτηση προς τον κύριο Μπουκ. Αναφέρετε την ευελιξία Και γνωρίζουμε, ακούσαμε και όλες, ότι για να διατηρηθεί η ευελιξία, για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιούμε ολική ενέργεια, πρέπει να υπάρχουν τεράστια αποθέματα ενέργειας. Αυτό μειώνει την ενεργειακή απόδοση αλλά από αυτά που είπατε, ότι δηλαδή 550 γραμμάρια ανά είναι το σύνηθες στη Γερμανία, υπάρχει ένα σχέδιο, μια πρόταση, η αιωλική ενέργεια να χρησιμοποιείται μαζί με την ενέργεια από φυσικό αέριο. 20 δηλαδή 30% αιωλικής ενέργειας και ανεμογεννήτριες που λειτουργούν με φυσικό αέριο. Αυτό θα παρέχει την αναγκαία ε, ευελιξία και την ενεργειακή απόδοση. Σας ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Μόρτεν Πέτερσεν έχει το λόγο τώρα. Εκπρόσω... Είναι εισηγητής της έκθεσης Acer. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ένα σχόλιο θα ήθελα να κάνω και μετά μια ερώτηση. Να σας ευχαριστήσω πρώτα για τις παρουσιάσεις σας. Ακούσαμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Ένα σχόλιο όμως έχω να κάνω για την παρουσίαση του ε, Δ. που τόνισε την σημασία των ε, δικτύων ενέργειας. Συμφωνώ πως είναι πολύ σημαντικά ιδιαίτερα ε, σε ό,τι αφορά τον κανονισμό ΕΑΣΑ. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ. Μία ερώτηση, λοιπόν, για τον κύριο Μπουκ και για την παρουσίασή του. Σε μία από τις διαφάνειές σας, ε, υπήρχαν πολλά στοιχεία, δεν είχα τα γυαλιά μου, δεν μπορούσα να διαβάσω. Ε, αυτό που είδα είναι ότι οι διαφάνειές ήταν φορτωμένες. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ που μας τις δώσατε και ε, τυπωμένες. Έχω λοιπόν μία ερώτηση σε σχέση με το πλαίσιο για τις ανανεώσιμες. Αναφέρεται ότι η εκτίμηση αντικτύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, αποκρύπτει τα ωφέλη των ανανεώσιμων και ε, παρουσιάζει το κόστος μεγαλύτερο από όσο είναι. Ε, θα ήθελα να μου σχολιάσετε αυτό το σημείο και θα με ενδιαφέρει να μάθω αν έχουν γίνει κάποιες σχετικές μελέτες που το αποδεικνύουν και που στηρίζουν του, τις εκτιμήσεις σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο εισηγητής για την ε, διακυβέρνηση, κύριος Τούρμας. Ευχαριστώ πολύ. Μία ερώτηση προς τον εκπρόσωπο της EX. Ποια είναι η σύνδεση ανάμεσα ε, στα προϊόντα μας, ε, μα μας είπατε για βραχή πρόθεσμα, για μακροπρόθεσμα και σε αυτό που ρώτησε και ο κύριος Σκάριντς ε, και στην αγορά, στο είδος της αγοράς που πρέπει να δημιουργήσουμε. Πώς πρέπει να είναι αυτή η αγορά με την αποθήκευση ενέργειας, ε, με τον ανοιχτό κύκλο, κλειστό κύκλο, ανεμογεννήτριες που λειτουργούν με φυσικό αέριο κτλ. Πού είναι η σύνδεση όλων αυτών με τις αγορές που θα ε, δούμε στην Ευρώπη. Και άλλη μια ερώτηση. Κύριε Μπουκ, πρόσφατα υπήρξαν δύο προτάσεις ε, για για... για αιωλική ενέργεια στην Ευρώπη. Η μία πρόταση ήταν για 55 ευρώ τη μεγαβατόρα και άλλη για περισσότερα. Η τεχνολογία αυτή δεν είναι κάτι καινούριο. Γιατί όμως υπάρχουν διαφορές στις τιμές, γιατί στην Πολωνία είναι πιο φθηνή η ενέργεια, είναι 40 ας πούμε, ευρώ την μεγαβατόρα από ό,τι στη Δανία. Οι χώρες αυτές δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη, ούτε η μία ούτε η άλλη. Πώς μπορούμε λοιπόν να εξηγήσουμε μια τόσο μεγάλη διαφορά τιμών και τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Γιατί αυτό δείχνει κάποια ανομαλία στις τιμές. Παρότι δηλαδή κάποια, η Πολωνία ας πούμε είναι χώρα με χαμηλότερο κόστος ζωής, η ενέργεια είναι πιο ακριβή. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Η κυρία Βέρνερ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δύο ερωτήσεις έχω προς τους προσκεκλημένους μία για, την, ε, για τις ζώνες τιμολόγησης και πώς αυτές ε, χωρίζονται. Πού βρίσκονται τα σύνορα ε, και θα έχουμε προβλήματα στην μετάβαση από τη μία ζώνη στην άλλη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα... Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μάλλον θα είναι αυτή που θα αποφασίσει που θα χωρίζονται, πώς θα χωρίζονται αυτές οι ζώνες που θα σταματάει μία και θα αρχίσει η άλλη. Εγώ θεωρώ πως αυτή η προσέγγιση είναι λάθος διότι με την πρόταση της Κομισιόν τα εθνικά μέτρα είναι αυτά που προτιμώνται για να ξεπεράσουν τα εμπόδια που θα δημιουργηθούν. Για παράδειγμα, η ε, ζώνη Γερμανίας και Αυστρίας ε, είναι η πιο ρευστή ζώνη στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Αγορά Ενέργειας και αυτό θα ήταν λοιπόν αντιπαραγωγικό γιατί θα έβαζε σε κίνδυνο τις άλλες ε, ζώνες τιμών. Μετά, η αξία του χαμένου ενεργειακού, ε, του χαμένου φορτίου. Αυτή είναι μια θεωρητική αξία, είναι μια εκτίμηση, ένας υπολογισμός ε, του κόστους της ενέργειας που θα χαθεί εάν γίνει κάποια διακοπή ρεύματο ή κάτι τέτοιο. Τα κράτη-μέλη όμως πρέπει να καθορίσουν αυτή την τιμή, τη θεωρητική τιμή, πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα έχουμε 27 διαφορετικές ε, τέτοιες ε, τιμές ε, χαμένης ενέργειας και, για, και πώς θα αποφύγουμε την στρέβλωση της αγοράς. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ρόιλ. Και εγώ έχω μια ερώτηση προς την Acer. Πολλέ φορέ έχω ζητήσει την Ευρωπαϊκή, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή απάντηση, αλλά δεν έχω πάρει. Γιατί δηλαδή η Acer να αποκτήσει ακόμα περισσότερες αρμοδιότητες. Ήδη υπάρχουν προβλήματα, θα δημιουργηθούν ακόμα περισσότερα. Μπορεί κάποιο να μου δείξει... Ε, το όφελος, μπορεί να μου δείξει κάποιο το, ότι χρειάζεται αυτή η ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της ΕΙΣΑ. Μετά, Υπάρχουν ήδη δυσκολίες να μεταφερθεί ενέργεια από τη μία χώρα στην άλλη, διασυνοριακά. Δηλαδή, στη Γερμανία, ας πούμε, πολύ δύσκολο να μεταφέρεις ενέργεια ε, από μια γειτονική χώρα. Δεν υπάρχει ετοιμότητα ακόμα. Γιατί, μήπως επειδή υπάρχει μια τεράστια ας πούμε εθνική οδός ε, ηλεκτρικής ενέργειας, ας το πούμε έτσι, ε, σε μια χώρα και όταν φτάνει στη Γερμανία χωρίζεται σε μικρά δρομάκια μήπως φταίει ότι τα δίκτυα δεν είναι κατάλληλα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μας δίνει κάποια συγκεκριμένη απάντηση. Όλα τα συμπεριλαμβάνει κάτω από το ναι πρέπει να δοθούν περισσότερες αρμοδιότητες στην ΕΣΑ. Μετά οι μηχανισμοί ε, ηλεκτροπαραγωγικών ικανοτήτων, οι, οι εκπομπές εκεί υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία της Κομισιόν βασίζονται σε μελέτες ή είναι όλα θεωρητικά. Ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφος Ντανίκα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Αν κατάλαβα καλά, όλες οι επιδοτήσεις για κάθε μορφή ενέργειας θα καταργηθούν. Είτε πρόκειται για ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, ε, για ορυκτά καύσιμα, πυρηνική, όλε οι επιδοτήσει θα καταργηθούν. Καλό αυτό, θα υπάρχουν επιδοτήσει μόνο για τι νέε τεχνολογίε. Όμω έχω ένα προβληματισμό, μία ερώτηση που θέλω να σα θέσω. Ίσως ο κύριος Παύλων θα μπορούσε να απαντήσει. Στη Ρουμανία είδαμε ότι ε, ένας ενδιάμεσος, μία offshore, αγόραζε 10 ευρώ την ενέργεια και την ε, μεταπολούσε στην αγορά. Η διαφορά από τα 10 στα 50 που πολλούσε, τα έβαζε στην τσέπη. Οι διασυνοριακές συναλλαγές πρέπει να γίνονται χωρίς καμία επιδότηση, αλλά με κάποιον φόρο τύπου ΦΠΑ. Μετά, ο μηχανισμός ε, ικανότητας, συγχωρητικότητας. Στη Ρουμανία το Γενάρη, για 10 μέρες, είχαμε ε, μείον 20 βαθμούς και με, με πολύ έντονους ανέμους, που σημαίνει ότι ουσιαστικά η, η θερμοκρασία πραγματικά ήταν κάτω από μείον 30. Προσπαθήσαμε να δανειστούμε από την Ευρωπαϊκή ε, Τράπεζα Επενδύσεων για να επεξεργαστούμε τις υποδομές μας, όμως τελευταία στιγμή δεν υπεγράφει η σύμβαση γιατί δεν πρόκειται για επένδυση που θα είχε σημαντική απόδοση. Και οι αρμόδιοι δεν μπορούσαν, για το έργο δεν μπορούσαν να αποδείξουν ότι όντω θα είχε ε, σημαντική απόδοση το έργο. Τι θα γίνει στην επόμενη χρονιά στη Ρουμανία. Εάν υπερβούμε το όριο των 550 μιλιγκράμμων που έχει οριστεί, τότε έχουμε πρόβλημα ε, σε ό,τι αφορά τις δικές μας, ε, τις δικούς μας ενεργειακούς πόρους. Ε, πρέπει να εισάγουμε από τους γειτονέ μας. Οι Ρώσοι που μας δίνουν μας είπαν λυπούμε, θα δεν μπορούμε να δώσουμε περισσότερο. Οπότε θα ανέβουν οι τιμές κατά 50%. Τι θα κάνουμε εμείς λοιπόν. Μετά θα ήθελα μια απάντηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, πρώτα απ' όλα μια παρατήρηση. Ο πρώτος ομιλητής ανέφερε ότι δεν πρέπει να ε, συγχέουμε τους ε, στόχους της ενεργειακής πολιτικής με την περιβαλλοντική πολιτική. Είναι δύο τελείως διαφορετικά ζητήματα, είπε τα οποία θα πρέπει να συζητήσουμε αλλού. Όμως, ο τρίτος ομιλητής είχε εντελώς διαφορετική στάση. Δεν ακούτε τη διερμηνία. Ωραία. Λοιπόν, είχατε μια πολύ διαφορετική προσέγγιση ότι η ενεργειακή πολιτική θα πρέπει ε, να υπάγεται πλήρως ε, στην ενεργειακή πολιτική. Το οποίο προκύπτει μάλλον και από το όνομα της, ε, του οργανισμού, το Energy Vende. Όμως έχουμε μια χώρα στην Ευρώπη που έχει πραγματικά πρωτοπόρο ρόλο σε όλη αυτή την ενεργειακή μετάβαση και από την εμπειρία αυτού του κράτους μέλους θα πρέπει να αντλήσουμε ορισμένα διδάγματα καθώς επεξεργαζόμαστε την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Και να σας ρωτήσω, από όσο ξέρω, όλοι αυτοί οι στόχοι της συνεργικής μετάβασης έρχονται ε, αντιμέτωποι με σημαντικές πρακτικές δυσκολίες. Μία από αυτές τις δυσκολίες είναι αυτό το απόθεμα, αυτό το backup που αναφέρθηκε προηγουμένως. Και υπάρχουν ε, προβλήματα εδώ στις υποδομές. Και η ενεργική μετάβαση δημιουργεί προβλήματα και από πλευρά γειτονικών χωρών που έχουν όλα ένα και μεγαλύτερα προβλήματα με την ενεργική πολιτική. Λοιπόν, θα ήθελα να ρωτήσω τον πρώτο μιλητή πώς αυτό συνδέεται με, την, αυτό που είπατε προηγουμένως ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει η επαρκή ολοκλήρωση στις ανανεώσιμες. Μπορείτε να μας δώσετε ορισμένα παραδείγματα. Πώς δηλαδή η δημιουργία τέτοιων ε, ζωνών υποβολής ενδιαφέροντος και προσφορών θα μπορούσε να ε, βοηθήσει στην τομέα των ε, ανανεώσιμων. Ευχαριστώ. Δύο θέματα θα ήθελα να θέσω. Το πρώτο είναι μια πραγματική απορία. Πώς θα πάμε από την κατάργηση των επιδοτήσεων προς μορφές ενέργειας όπως είναι οι, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην ομαλοποίηση της αγοράς. Ποιο μηχανισμό ή ποιοι μηχανισμοί προτείνονται ώστε να μην καταστραφούν οι επενδυτέ σε αυτέ τι μορφέ ενέργεια που έχουν ήδη κλείσει συμφωνίε σε υψηλέ τιμέ και συγχρόνω να μην υποστούν ζημιά τα κράτη-μέλη. Το δεύτερο αφορά στην ασφάλεια. Ξέρετε υπάρχουν κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα οποία δεν περιβάλλονται από άλλα κράτη-μέλη μόνο. Και ένα παράδειγμα είναι η δική μου χώρα, η Ελλάδα, που περιβαλλέται από υποψήφιου χώρε, αλλά και από χώρε με τι οποίε υπάρχει κάποια στιγμή ένταση, όπω είναι η Τουρκία. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω πώς μπορείτε να, να σκεφτείτε, πώς μπορείτε να σχεδιάσετε ένα μηχανισμό διασυνοριακής υποστήριξης ώστε να υπάρχει η ασφάλεια στην παροχή χωρίς ταυτόχρονα η ίδια η, η, ενεργειακή επάρκεια τέτοιων χωρών να μπαίνει σε κίνδυνο. Σας ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Χάμς. Yeah. You are on the list. You are on the list of speakers. Thank you. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να υπογραμμίσω ότι όλο αυτό το πακέτο, το χειμερινό πακέτο είναι πολύ σημαντικό να το δούμε ταυτόχρονα με, τη, το θέμα με την θέσπιση στόχων για το κλίμα, για την ενεργειακή μας πολιτική. Αυτό το χειμερινό λοιπόν πακέτο πρέπει να ε, έχει ως στόχο την ε, αποδέσμευση της, ενέργειας, της ενεργειακής μας παροχής από τον άνθρακα. Γι' αυτό θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μπουκ ποια είναι η αιτιολογία για τις επιδόσεις εκπομπών, για το emission performance που μας είπατε. Εγώ θεωρώ απαραίτητο, αναγκαίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να προτείνει κάτι τέτοιο όπως και έκανε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ένστ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα αναφερθώ σε δύο θέματα. Καταρχάς μιλάμε πολύ για καθαρή ενέργεια και για ε, το πώς θα καθοριστούν οι τιμές, πώς θα ε, δημιουργήσουμε περισσότερες ανανεώσιμες, ε, πώς οι τιμές θα είναι λογικές. Όμως Ας μην ξεχνάμε και την ενεργειακή ένδυα. Ιδιαίτερα σε πολλές χώρες της Νότιας, Νοτιοανατολικής Ευρώπης υπάρχει αυτό το ε, πρόβλημα και είναι αρκετά έντονο. Πώς μπορούμε λοιπόν να συνδέσουμε αυτόν τον στόχο της καθαρής ενέργειας δηλαδή και της ε, ενεργειακής ένδυας που υπάρχει σε κάποια κράτη-μέλη που πολλές φορές ε, για να ζεστάνουν τα σπίτια τους χρησιμοποιούν ακατάλληλες ε, μεθόδους, ακατάλληλους τρόπους. Πώς μπορούμε λοιπόν να αλλάξουμε τα πράγματα προς το καλύτερο. Και μετά κάτι άλλο για τις ανανεώσιμες. Τους τελευταίους μήνες πάντα ε, συζητάμε το θέμα της αποθήκευσης ενέργειας, των, των αποθεμάτων, όμως από ό,τι καταλαβαίνω δεν είμαστε ευχαριστημένοι με το πώς έχουν τα πράγματα τώρα. Με το νομοθετικό πλαίσιο χρειάζεται ένα πιο στιβαρό ε, πλαίσιο έτσι ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση. Εσείς θεωρείτε πως είναι επαρκές το εφισταμένο πλαίσιο, οι προτάσεις που έχουν γίνει. Μετά, εντάξει, ακούμε πολύ για καθαρή ενέργεια, ότι θέλουμε αποδέσμευση από άνθρακα κτλ. κτλ, κτλ. Ε, τι κάνουμε όμως στην πράξη, στηρίζουμε κάποιες ε, προτάσεις, κάποιες ε, ενέργειες, δράσεις. Ο κύριος Κέλλη έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τους ομιλητές. Εγώ είμαι από την Ιρλανδία και βεβαίως Έχουμε αναλάβει δεσμεύσει σε ό,τι αφορά την κλιματική αλλαγή και την εισαγωγή περισσότερων ανανεώσιμων πηγών ενέργεια στο σύστημα. Όμω υπάρχει μια δυσκολία τώρα που συνδέεται με το Brexit. Δεν θα συνδεόμαστε πλέον με την ευρωπαϊκή επικράτεια. Υπάρχει λοιπόν και μια πρόταση να υπάρξει ένας, ε, μια υποδομή διασύνδεσης ε, ηλεκτρικής ενέργειας που είναι Βέβαια κάτι πολύ σημαντικό, σίγουρα όμως και πολύ δαπανηρό. Υπό ιδανικές συνθήκες η Ευρώπη θα είχε αυτή τη διασύνδεση. Αυτό θα ήταν τμήμα της Ενεργειακής Ένωσης. Όμως, πώς μπορεί να γίνει αυτό στην πράξη και είναι κάτι το οποίο μα παίρνει οικονομικά. Δεύτερον, αυτό που έθιξαν συνάδελφοι ε, για το backup, το απόθεμα ε, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αν συνεχιστεί ε, η έρευνα και έχουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όχι μόνο τις γνωστές, αιωλική και ηλιακή, αλλά για παράδειγμα, πέρσι, συνάδελφοι ήταν στη δική μου εκλογική περιφέρεια, όπου γίνεται ε, έρευνα ε, και σε νέες μορφές ε, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που κάποια στιγμή θα γίνουν πραγματικότητα όπως και η ολική Κυριακή σήμερα. Αν είχαμε λοιπόν αυτές τις υποδομές διασύνδεσης, ίσως αντί να έχουμε ορυκτά καύσιμα ως ε, ε, backup στα ανανεώσιμα, ίσως να συνέβαινε το αντίθετο. Οι ανανεώσιμες να ήταν δηλαδή ε, λύση ανάγκης ε, για τις ορυκτές. Θα είχαμε και τα δύο δηλαδή. Μήπως όμως θα πρέπει να δώσουμε έτσι προτεραιότητα στην διασύνδεση της Ευρώπης, να δημιουργήσουμε μια πραγματική ενεργειακή ένωση για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και μετά όλα αυτά για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα γίνουν πιο εφικτά and, uh, Παρακαλώ σχόλια και απαντήσεις. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Εφόσον υπήρξαν πολλές ε, διαφορετικές θεματικές ενότητες που έθιξαν ε, συνάδελφοι, αρχικά να σας ευχαριστήσω για τις ερωτήσεις σας. Νομίζω ότι πραγματικά είναι κέρυες οι παρεμβάσεις σας. Κύριε Κάριντς, κατά κάποιον τρόπο είπατε ότι θα έπρεπε να έχουμε ε, η ικανότητα τα, και τα αποθέματά μας θα πρέπει να είναι ένα προς ένα σε σχέση με τους ενεργειακούς μας πόρους. Από αναλυτικής άποψης, εμείς δεν ε, συμμεριζόμαστε αυτή την άποψη αν δείτε ορισμένα τα κράτη-μέλη που έχουν πολύ υψηλά μερίδια ανανεώσιμων ήδη στον ενεργειακό τους μείγμα σήμερα, όπως η Ιρλανδία, η Δανία, εκεί δεν υπάρχει αυτός ο λόγος ένα προς έναν σε ό,τι αφορά την ε, ικανότητα που χρειάζονται αυτά τα κράτη-μέλη. Μάλιστα, ε, υπάρχουν μελέτες ε, που εξετάζουν το μέλλον μακροπρόθεσμα και βλέπουν το ζήτημα της αποθήκευσης. Και ξέρουμε ότι αυτό θα πάρει χρόνο. αλλά σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό ε, σε σχέση με σήμερα. Είναι σημαντικό λοιπόν πόσα από θέματα χρειαζόμαστε, είναι υπεραπλησιαστικό να λέμε ότι ο λόγος θα είναι ένα προς έναν. Με τα χαράς ε, να το συζητήσουμε και διμερώς, αν θέλετε. Επίσης, ήθελα να σταθώ σε κάτι που ανέφεραν πολλοί ε, ομιλητές για τα 550 γραμμάρια, αυτό το όριο που έχει τεθεί στις εκπομπές. Είπατε ότι αυτό συνδέεται με μια γερμανική συζήτηση, κύριε Κυριακ. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτή την ε, άποψη. Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όταν έκανε αυτή την πρόταση, ρητός ε, ξεκαθάρισε και αυτό αντανακλά και όλη την προσέγγιση της Ενεργικής Ένωσης, δηλαδή ότι θέλουμε να έχουμε μια συνέπεια, μια ολιστική προσέγγιση και ότι έτσι θα πρέπει να έχουμε κατά νου τους ε, στόχους για την κλιματική αλλαγή όταν ε, θέλουμε να σχεδιάσουμε την ε, αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας. Ήδη από το 2013 έχει αρχίσει να ασχολείται με αυτό το ζήτημα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Δεν στηρίζονται προγράμματα τα οποία δεν συμμορφούνται με το όριο αυτό των 550 γραμμαρίων. Ήδη λοιπόν αυτό εφαρμόζεται από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θεωρώ ότι η πολιτική της εξάλληψης ε, των ρηπαρών ουσιών για το περιβάλλον είναι μια μακροχρόνια διαδικασία. Αυτό το πρότυπο των 550 ε, γραμμαρίων ισχύει μόνο ε, στο μηχανισμό ικανότητας για τον οποίο λαμβάνουμε επιδότηση. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν αυτό πληρεί αυτό το κριτήριο που προανέφερα. Και ότι βεβαίως δεν ε, επιδοτούμε ε, πολιτικές και μεθόδους που ρηπαίνουν το περιβάλλον. Κύριε Τούρμες, ε, ρωτήσατε ποια είναι η διαφορά ε, μεταξύ Δανίας και Πολωνίας και για την τιμή της ενέργειας. Αυτό συνδέεται και με το προηγούμενο ερώτημα του κόστους. Γιατί δηλαδή το ρίσκο μεταφράζεται σε κόστος. Το είπατε και εσείς κύριε Κάρινς. Ίσως να μην το εξήγησα αρκετά διεξοδικά. Από πλευρά επενδυτή, οι επενδύσεις αυτές για τις ανανεώσιμες είναι Ε, υψηλής ε, απέτησης ε, επενδύσεων και κεφαλαίων. Επομένω, είναι πολύ υψηλό το κόστος και έτσι είναι πολύ μεγαλύτερη η εξάρτηση από μια σταθερή προοπτική μελλοντικά. Πολιτικό, προσκήνιο, οικονομικό, υποδομές και το Και από πλευράς ε, εξάντε προσδοκιών, αυτό συνδέεται και με το τέλος ε, ρίσκου. Το risk premium λοιπόν προστίθεται στο κόστος της επένδυσης. Και τώρα κύριε Τούρμες, αν δείτε τον ε, χάρτη της Ευρώπης αυτή τη στιγμή, έχουμε διαφορετικό κόστος κεφαλαίου για επενδύσεις ανανεώσιμων στα διάφορα και γιατί συμβαίνει αυτό. Αυτό μπορεί να συνδέεται με τις διαφορετικές επιδόσεις του ρυθμιστικού περιβάλλοντος στα επιμέρους, κράτους, στα επιμέρους κράτη-μέλη. Ή μπορεί να ισχύει και με την ίδια την ε, χώρα και γενικότερα τους κινδύνους ε, της οικονομίας σε αυτή τη χώρα. Επομένω, η ίδια επένδυση φωτοβολταϊκών ε, κοστίζει περισσότερο αυτή τη στιγμή στην Πολωνία από ό,τι στη Δανία. Με τη δική μας ανάλυση λοιπόν, εξετάζοντας έναν ευρωπαϊκό δεσμευτικό στόχο, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στο πακέτο. Και στην πρόταση ΑΠΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάρχει μια πρόταση, και μια βάση συζήτησης όπου θα πρέπει να εξετάσει το κόστος του κεφαλαίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε κάθε κράτος μέλος. Νομίζω τα απάντησα. Ναι, βεβαίω, θα δώσουμε το λόγο στου υπόλοιπου ομιλητέ, Κύριε Μπουκ. Ενεργή Βέντε. Παρακαλώ, κυρία Νή. Μου ζητήθηκε να απαντήσω σε τέσσερις ερωτήσεις. Κύριε Κάρινς, για τους μηχανισμούς χωρτικότητας. Ε, δεν μπορούμε ε, να... Δεν μπορώ να απαντήσω έτσι με άσπρο ή μαύρο, αλλά πραγματικά υπάρχουν πολλά κουτάκια τα οποία πρέπει να ε, διαγράψουμε ότι δεν πρέπει να κοιτάμε μόνο την παραγωγή ενέργειας, αλλά όλες τις άλλες δυνατότητες για ενεργειακή απόδοση. Χρειάζεται λοιπόν να σημειώσουμε και το, ε, το login του άνθρακα, έτσι ώστε να γίνει η ενεργειακή μετάβαση. Για να γίνει όμως η ενεργειακή μετάβαση πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τις ε, διασυνδέσεις περιφερειακές, ε, διακρατικές και να υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές για να γίνει αυτό. Ε, και αυτός ο μεταβατικός χαρακτήρας σημαίνει ότι μετά από αυτήν την εκτίμηση για την επάρκεια ενέργειας ε, πρέπει να ακολουθήσει και ένα ενεργό σύστημα ενεργειακής διαχείρισης. Να χρησιμοποιήσουμε δηλαδή τις ευκαιρίες που μας δίνει η ψηφιακή ενία αγορά για να βελτιστοποιήσουμε ένα σύστημα που ο πελάτης ε, θα ε, καθορίζει τις εξελίξεις. Αυτή είναι η νέα φάση της ενεργειακής μετάβασης. Εάν μπορούμε λοιπόν στο κουτάκι να σημειώσουμε ναι, τότε θα έχουμε κάνει καλά τη δουλειά μας. Μετά η κυρία Βέρνερ έκανα μια ερώτηση σχετικά με το πώς ε, καθορίζονται αυτές οι ζώνες τιμολόγησης. Είναι σαφές ότι για ορισμένα μέρη της Ευρώπης αυτό ο διαχωρισμός είναι καταστροφικός και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Όταν θέλεις να ενώσεις ε, με αυτόν τον τρόπο κάνεις το ακριβώς αντίθετο υπάρχουν πολλά ε, σημεία που είναι προβληματικά, πολλές ελλείψεις και η έλλειψη για παράδειγμα ενός ε, δικτύου που να ενώνει με το Νότο είναι ε, ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή η, η δυνατότητες σύνδεσης Γερμανίας και Δανίας χρησιμοποιούνται κατά 60%. Στο νότιο κομμάτι όμω, υπάρχουν προβλήματα και υπάρχει πρόβλημα στη σύνδεση βόρειας και νότιας Γερμανίας ενεργειακά. Πρέπει λοιπόν να βρούμε ποια θα είναι η καλύτερη δυνατή λύση. Και ε, δυστυχώ προ το παρόν η καλύτερη δυνατή λύση φαίνεται ότι είναι αυτό ο διαχωρισμό σε δύο διαφορετικέ ζώνε τη ίδια χώρα αυτή τη στιγμή καταρτίζεται μία μελέτη για τις ζώνες τιμολόγησης, αλλά στο τέλος η απόφαση δεν θα είναι δική μας, ούτε των επιστημόνων θα είναι πολιτική. Κύριε Ρόιλ, ζητήσατε να σας απαντήσω γιατί χρειαζόμαστε μένα γιατί διατή Acer, γιατί χρειάζονται ή μήπως είναι καλύτερο να δημιουργηθούν ισχυρότερα και καλύτερα δίκτυα. Και τα δύο θα σας απαντήσω εγώ. Πρέπει, στη, όπως θα δείτε και στην μελέτη μας, να δούμε τις ανάγκες που έχουμε σήμερα. Εάν θέλουμε πραγματικά να υπάρξει μία ενιαία αγορά ενέργειας, χρειάζεται καλύτερη νομοθεσία, ένα βελτιστοποιημένο σύστημα και αυτό που μάθαμε από την εμπειρία του ΕΣΕΡ 2009 ε, μας δίδαξε ότι όταν δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε κάποια αδιέξοδα λόγω εθνικών συμφερόντων, χρειάζεται καλύτερη νομοθεσία και να επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας σε άλλους τομείς. Γι' αυτό χρειάζεται καλύτερη εποπτεία και έλεγχος. Μετά, Δύο φορές με ρώτησε ο κύριος Νίκα από τη Ρουμανία. Υπήρχαμε και μια ερώτηση από την ε, Ελλάδα για την ενεργειακή, ε, την ασφάλεια του εφοδιασμού, του ενεργειακού εφοδιασμού. Ε, υπάρχουν και περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Τον Ιανουάριο μείον 20 βαθμούς έφτασε στην Ελλάδα. Α, λέτε κάθε χρόνο συμβαίνει αυτό. Ζητώ συγγνώμη τότε, αλλά ε, τα στοιχεία που είδαμε εμεί, ε, τα πιθανά σενάρια, ε, μας έδειξαν ότι αυτή είναι συνήθιστη περίπτωση τόσο χαμηλών θερμοκρασιών. Είδαμε όμως ότι κάθε χώρα προσπάθησε να λύσει το πρόβλημα μόνη της σε τέτοιες περιπτώσεις και η λύση θεωρούμε πως είναι η περιφερειακή συνεργασία. Αυτό όμως εξαρτάται από τη διακυβέρνηση, από τις ε, αρχές, από την ηγεσία και αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να κοιτάξουμε αυτά τα θέματα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης με την Ομάδα Συντονισμού Ηλεκτρικής Ενέργειας έτσι ώστε να ε, λυθούν τα προβλήματα των πολιτών αυτών των χωρών. Τέλος, ε, αναφέρθηκε η ενεργειακή ένδυα και τι κάνουμε στην περίπτωση χωρών που οι πολίτες τους δεν μπορούν να, ε, να και χρησιμοποιούν ξύλα ή άλλους τρόπους να ζεστάνουν τα σπίτια τους. Αυτό είναι κάτι που γνωρίζουμε εδώ και αρκετό καιρό, ένα γνωστό θέμα και η απάντηση μπορεί να είναι να δώσουμε τη δυνατότητα στους ανθρώπους να κάνουν πράγματα. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, έχουμε το, την... Ε, κάτι ε, προγράμματα την, ε, που στηρίζονται από την τράπεζα KFW. Έχουμε κάποια δάνεια με χαμηλό επιτόκιο, κάποιες επιχορηγήσεις για ε, να μονώσουν οι πολίτες στα σπίτια τους και προσπαθήσουμε να, προσπαθούμε να βοηθήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Ε, δυστυχώς όμως οι ίδιες λύσεις δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε όλες τις περιπτώσεις υπάρχουν ορισμένες ε, χώρες όπου οι τιμές άλλαξαν και στρεβλώθηκαν τεχνητά. Ευχαριστώ πολύ. Την κυρία Ρης. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Πάολουν για τα τελευταία σχόλια αυτού του πάνελ. Σα ευχαριστώ. Η ερώτηση που μου θέσατε είναι κατά πόσο οι αγορέ μπορούν να κρατήσουν την ασφάλεια ανεφοδιασμού. Ναι, μια τέτοια ενιαία αγορά θα μπορούσε όντω να στηρίξει την ασφάλεια ανεφοδιασμού και ε, να έχει τα αντίστοιχα επενδυτικά σήματα καθώς και τα έσοδα για να χρηματοδοτήσει οι επενδύσει. Σε ένα τέτοιο σενάριο φυσικά το πραγματικό επίπεδο ασφάλεια ανεφοδιασμού είναι το οικονομικό αποτέλεσμα τη αγορά, δηλαδή η, η αγορά αποκαλύπτει την πραγματική αξία. Και δεν είναι βέβαιο ότι αυτό το επίπεδο ασφάλειας ε, ανεφοδιασμού θα είναι το ίδιο με το σημερινό ή υψηλότερο. Εάν θέλουμε να πετύχουμε ένα συγκεκριμένο επίπεδο ασφάλειας ανεφοδιασμού που να είναι πάνω από το οικονομικό αποτέλεσμα της αγοράς, τότε θα χρειάζονται πλέον επενδύσεις. Ε, και θα χρειαστούν και επιπλέον μηχανισμοί χωρητικότητας ή μηχανισμών. Και άλλα παραδείγματα μπορεί να είναι, ας πούμε, η προσωρινή προσωρινή ε, πλέγματος, όπου έχουμε ε, περιορισμό της ε, παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Χρειάζονται λοιπόν προγράμματα στήριξης επιπλέον που θα πρέπει να σχεδιαστούν με τέτοιο τρόπο ώστε να μην τρευλώνουν τις τιμές της αγοράς. Ε, αναφέρθηκε και άλλη μια ερώτηση στην ε, δυνατότητες της αγοράς και πώς αντιμετωπίζουμε την κατάσταση όπου ισχύουν διαφορετικοί κανόνες από τις δύο πλευρές των συνόρων. Ακριβώς περί αυτού πρόκειται. Αν η δεν υπάρξει συντονισμός, τότε υπάρχει αστρέβλωση της αγοράς στα σύνορα. Γι' αυτό και είναι τόσο σημαντικό να έχουμε κοινά κριτήρια και να έχουμε μια σωστή εξολόγηση από την αρχή για το κατά πόσο ο μηχανισμός ε, δυνατοτήτων χρειάζεται, λαμβάνοντας υπόψη και τη διασυνοριακή, τις συνοριακές δυνατότητες των δύο όμορων χωρών ή κατά πόσο άλλες γειτονικέ χώρες μπορούν να συμβάλλουν στην ασφάλεια ανεφοδιασμού και λίγο πιο πέρα από τα σύνορα. Τώρα τέθηκε το θέμα της ευελιξίας. Τι είδους αγορές χρειαζόμαστε δηλαδή στο μέλλον για να μπορέσουμε να εσωματώσουμε τις νέες ε, ανάγκες. Δεν είναι είτε το ένα είτε το άλλο. Όλα αυτά μπορούν μαζί να συμβάλλουν στην ευελιξία και στην ασφάλεια ανεφοδιασμού να δώσω ένα παράδειγμα για το πώς λειτουργεί αυτό στην πράξη και μιλώ για την αγορά του IPEX Spot που είναι η πιο βραχυπρόθεσμη ρευστή ε, αγορά, δηλαδή οι συμβάσεις των 15, 15 λεπτες ή 30 λεπτες που μπορεί κανείς να εμπορευθεί αμέσως πριν την παράδοση. Έτσι υπάρχει και πραγματική ευελιξία στην αγορά. 30 λεπτά δηλαδή πριν από την παράδοση μπορούν όλοι οι μετέχοντες στην αγορά να πουλούν ή να αγοράζουν πραγματική ενέργεια στην αγορά. Πολύ σημαντική πηγή ευελιξία και πάει χέρι-χέρι με τους πραγματικούς παίχτες ε, όπως τους ε, φορείς αποθήκευσης, ε, τους παρόχου όσου έχουν ευελιξία στο χαρτοφυλάκιό του, μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτέ τι αγορέ ώστε τη δική του ευελιξία να τη διαθέσουν στου άλλου που τη χρειάζονται. Και όσοι περισσότεροι συμμετέχουν σε αυτό το σύστημα τόσο το καλύτερο. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μεγάλε αγορέ, Αλλά και οι αγορέ. futures το συμβάλλουν σε αυτό. Έχουμε σχεδιάσει ε, προϊόντα που τα ονομάζουμε Cup of Futures, που ακριβώς έχουν σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες ευελιξίας των φορέων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η βραχυπρόθεσμη αγορά είναι η πραγματική, όπου μπορεί κανείς να πουλήσει και να αγοράσει ηλεκτρισμό πολύ γρήγορα. Βέβαια, εκεί μπορεί να υπάρξουν διακοιμάσεις τιμών, όταν ας πούμε επιγόντως χρειάζομαι να αγοράσω ενέργεια, ε, πολύ βραχυπρόθεσμα, τότε η τιμή θα μπορεί να είναι πολύ ψηλότερη. Αν θέλω να αποφύγω αυτό το κίνδυνο, πρέπει να χρησιμοποιήσω τα εργαλεία στη μακροπρόθεσμη αγορά και να προσπαθήσω να έχω έτσι μια μεγαλύτερη ασφάλεια. Άρα, ο συνδυασμό όλων αυτών ε, παίζει ρόλο. Και αν δούμε τη γερμανοαυστριακή αγορά που, παίζει, που είναι πρωτοπόρα σε αυτό το τομέα, μπορούμε στην πράξη να δούμε πώ λειτουργεί το σύστημα. Αυτό που περιορίζει αυτή την αγορά είναι το ρυθμιστικό πλαίσιο, γιατί ακριβώ δεν δίνει κίνητρα ε, στους φορείς που ενδιαφέρονται για αυτά τα και του οποίου οποίους στοχεύουμε εμεί με αυτά τα προϊόντα να, να, να συμμετέχουν. Προσπαθούμε να ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα και είμαστε βέβαιοι ότι αυτό θα παίξει μεγαλύτερο ρόλο στο μέλλον. Uh, Well, if I may mm, uh, question, uh, if... Uh, Any Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, δεν νομίζω πως έμεινε κάποια αναπάντητη ερώτηση από τους προσκεκλημένους. Δεν βλέπω αντιδράσεις. Νομίζω πως απαντήσετε λοιπόν και καλύψατε όλα τα ερωτήματα. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν όλους τους ομιλητές για τις ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις σας, για τις ερωτήσεις, απαντήσεις. 27 ερωτήσεις, αν δεν κάνω λάθος. Και είναι εκπληκτικό που τις απαντήσατε τόσο γρήγορα. Και περνάμε τώρα στο δεύτερο μέρος της ακρόασής μας, το πώς θα ενταχθούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην αγορά ενέργειας, οι ευκαιρίες και τα εμπόδια. Θα ήθελα λοιπόν να αρχίσω με τον πρώτο προσκεκλημένο, να έρθει στο Προεδρείο για να αρχίσουμε ο πρώτος προσκεκλημένος είναι ο κύριος Χωσέ Ντονός, ο Γενικός Διευθυντής της UNEF, του... Ε, της, Ένωσης, ε, της Ισπανικής Ένωσης Φωτοβολταϊκών. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα προσθήκη στην ακρόασή μας, διότι ο κύριος Ντονόσο, Γενικός Διευθυντής, εκπροσωπεί την αγορά φωτοβολταϊκών στην Ισπανία. Και νομίζουμε πως υπάρχει πολύ μέλλον. Έχετε το λόγο. Okay. Any language you wish, 23 to your disposal. No, doesn't matter, but okay, the Spanish okay, will be more, more quick. Sorry. Okay, I, sorry for to pasar. Is it okay? Para pasar, for to go hit. Next to you. Okay. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα να παρουσιάσω ε, με τις απόψεις μας ε, σε αυτό το βήμα και θα προχωρήσω άμεσα στο θέμα. Τα τελευταία χρόνια είδαμε εντυπωσιακή μείωση στο κόστος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας παγκοσμίως, ιδιαίτερα Έχουμε μείωση 85% τα τελευταία χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι η ανανεώσιμη ενέργεια όχι μόνο είναι καθαρή, αλλά είναι και προσιτή. Τα εμπόδια στην ολοκλήρωση των ανανεώσιμων ε, στην αγορά εξακολουθούν να υπάρχουν. Το πρώτο είναι η έλλειψη νομικής βεβαιότητας και είναι πολύ σημαντικό η οδηγία που συζητάτε αυτές τις μέρες στο Κοινοβούλιο να αποκαταστήσει την κατάσταση. Η έλλειψη εμπιστοσύνη στην αγορά και στις εθνικές κυβερνήσεις μόνο μπορεί να διορθωθεί από την Κομισιόν και έτσι θα αποκατασταθεί η, θα αποκατασταθεί η νομική βεβαιότητα και γιατί περισσότερο κίνδυνο σημαίνει ψηλότερη τιμή. Τώρα, το, η τιμή, η τιμολόγηση. Θα θέλαμε να είμαστε μέσα στην αγορά, θα θέλαμε να συμμετέχουμε στην αγορά, αλλά το πρόβλημα είναι ότι οι αγορές δεν είναι οι ίδιες. Ο σχεδιασμός αυτής της αγοράς που ισχύει σήμερα είναι προ κονταετίας. Ο βασικός δηλαδή παράγοντας στην αγορά είναι η πηγή της ενέργειας που έχουμε εισάγει με μεταβλητό κόστος. Όμως οι ανανεώσιμες δεν έχουν μεταβλητό κόστος, οπότε υπάρχει μεγάλη αντίφαση που είναι η εξής. Εάν θέλουμε να τηρήσουμε τους στόχους του Παρισιού, κάθε χρόνο θα πρέπει να έχουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εισάγουμε την ηλεκτρισμό σε μηδενική τιμή και έχουμε μια αγορά όπου το σήμα είναι το περιθωριακό κόστος. Πρέπει δηλαδή να ξανασκεφτούμε το σύστημα της αγοράς. Στόχος θα πρέπει να είναι να δημιουργήσουμε μια νέα αγορά που θα συμφωνεί με την πραγματικότητα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Να σχεδιαστεί δηλαδή η αγορά με τρόπο ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί στην πραγματικότητα. Έπειτα. Δεν υπάρχει σαφής δρόμος για την οδηγία της ε, του άνθρακα όταν ο στόχος είναι μόνο 27% και τον έχουμε φτάσει χωρίς καμία ιδιαίτερη προσπάθεια, δεν σημαίνει αυτό πως υπάρχει πραγματική προθυμία από τις εθνικές κυβερνήσεις να προχωρήσουν το δρόμο των στόχων του Παρισιού. Ενώ ταυτόχρονα δεν θέλουν οι κυβερνήσεις να αναλάβουν εθνικές δεσμεύσεις. Αν θέλαμε να πάμε στο Παρίσι και να αυξήσουμε σε ένα πραγματικό στόχο αυτό το 27% που θα έδινε μήνυμα προς την αγορά ότι η προθυμία, ότι η βούληση των κυβερνήσεων είναι να τηρήσουν αυτές τις συμφωνίες, τότε θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε την βιομηχανία και την τεχνολογική βιομηχανία στην Ευρώπη να επενδύσει με εμπιστοσύνη στο μέλλον και να ε, κατακτήσει την ηγετική θέση που πρέπει να έχει η Ευρώπη σε παγκόσμιο επίπεδο στα θέματα της ενέργειας. Εφόσον δεν υπάρχει πραγματική βούληση για τη δημιουργία πιο καθαρής ενέργειας, θα είναι πολύ δύσκολο να αναπτυχθεί μια σημαντική αγορά για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι ανανεώσιμες παρουσιάζουν ευκαιρίες, μείωση του κόστους, δηλαδή μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα για τη βιομηχανία μας, συμβάλλουν κατά των κλιματικών αλλαγών, πρωτοπορία της Ευρώπης σε βιομηχανικό και τεχνολογικό επίπεδο, απασχόληση, δημιουργία μάλλον θέσεων απασχόλησης και νέες τεχνολογικές εξελίξεις στην οικοδόμηση αυτής της νέας αγοράς. και έτσι θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα το... Ε, ε, ε, αγορά ηλεκτρισμού όπως τη φανταζόμαστε. Όμως, για να δοθεί περισσότερη ισχύ στους καταναλωτές, πάλι έχουμε να αντιμετωπίσουμε εμπόδια. Κάθε, κάθε χρόνο βλέπουμε την ανόρθωση οικονομικών φραγμών για την κατανάλωση, την αυτοκατανάλωση. Είναι δικαίωμα που πρέπει να έχει ο καταναλωτής όταν έχει παραπάνω παραγωγή και μπορεί να εισάγει την παραπάνω αυτή η παραγωγή στο πλέγμα. Αλλά δεν πρέπει να χρεώνεται όταν χρησιμοποιεί τον ηλεκτρισμό εντός της οικία του. Γιατί αυτό δεν έχει γίνει ποτέ στην ιστορία της οικονομίας. Κάποιος να πληρώνει, να χρεώνεται για κάτι που ο ίδιος έχει κατασκευάσει και καταναλώνει. And every time there is more establishment of more administrative barriers Τώρα, Περισσότερα διοικητικοί φραγμοί επίση θεσπίζονται. Πρέπει όμως να καταργηθούν. Χρειαζόμαστε σύντομες διοικητικές διαδικασίες συμπεφωνημένες και αντίστοιχες με το πραγματικό μέγεθος της ε, παραγωγής. Φραγμή τώρα στην αποθήκευση. να μπορέσουμε να επενδύσουμε στην αποθήκευση και στο μέλλον θα δούμε ότι το σύστημα αποθήκευσης θα μπορεί να σταθεί σε ανταγωνιστικές τιμές στην αγορά. Επίσης χρειάζεται προσαρμογή των περιβαλλοντικών ε, ρυθμίσεων για την ε, αυτοκατανάλωση ώστε να μην ορθώνονται περαιτέρω φράγμοι. Ε, πρέπει από την πλευρά μας να μπορέσουμε να δουλέψουμε περισσότερο για την ολοκλήρωση των κτηρίων, για να μπορέσουμε να σεβαστούμε και την αισθητική των πόλεων μας. Έχουμε μια τεράστια ευκαιρία οι ανανεώσιμες δεν είναι μόνο ο τρόπος για καθαρή ενέργεια, αλλά και για προσιτή και ανταγωνιστική ενέργεια. Σας ευχαριστώ πολύ. For Σας ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Αρνό Σαπερόν αντιπρόεδρο της ΕΦΕΣ της, το ε, ΤΑΛ, μεγαλύτερου ομίλου φυσικού αερίου και πετρελαίου και ηγετική φυσιονομία στις, στις ανανεώσιμες. Ε, η Total δράση 123 χώρες, έχει 100.000 υπαλλήλους, είναι ένας τεράστιος αριθμός αυτός, πολλές δραστηριότητες. Έχετε αμέσως το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, εξότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, κύριε και κύριοι. Σας ευχαριστώ που μας κάνατε αυτή την εισαγωγή. Εγώ θα σας πω αυτά που είναι λιγότερο γνωστά, πέραν τις δραστηριότητε μας ε, στο φυσικό αέριο, στο πετρέλαιο και στην ε, ηλιακή ενέργεια. Είμαστε και πολύ μεγάλος παίκτη αυτή τη στιγμή ε, στις μπαταρίες, στους ισορρευτές, με την απόκτηση της SAFT πέρυσι. Ε, αλλά και στην ε, Χονδρική Κυλιανική ε, και συγκεκριμένα στο Βέλγιο με τη Λαμπυρίς. Έχουμε 4 εκατομμύρια καταναλωτές μέχρι σήμερα και 2 εκατομμύρια αυτών είναι στην Αφρική. Είναι με στρατηγική εδράζεται σε τρεις πυλώνες. Βελτίωση του ενεργικού μας μείγματος, ανάπτυξη των ΑΠΕ γιατί ξέρουμε ότι όλα αυτά αποτελούν, θα αποτελούν τα 20% του χαρτοφυλακίου της Total μέσα στην επόμενη 20 ετία και θέλουμε να γίνουμε ένας από τους τρεις ε, βασικούς φορείς παγκοσμίω στην ηλιακή ενέργεια. Ε, θέλουμε να προσθέσουμε και την ε, αποθήκευση ενέργειας στις δραστηριότητές μας, δραστηριότητές μας, αλλά και την ανάπτυξη της βιοτεχνολογίας. Θέλουμε να βελτιώσουμε την ενεργειακή απόδοση, προωθώντας την υπεύθυνη κατανάλωση ενέργειας και από τους καταναλωτές μας. Ας ξεκινήσω πρώτα από την τιμολόγηση του άνθρακα, που είναι πολύ σημαντικό στοιχείο της ενεργειακής μετάβασης. Θα συζητηθεί σύντομα στον τριμερή διάλογο για την αναθεώρηση του ETS. Είναι από τα κρίσιμη σημασία στοιχεία. Πράγματα, πραγματί δεν μπορούμε να ε, διατηρήσουμε αυτή την τιμολόγηση των 5 ευρώ τόνο. Ο μηχανισμός ETS ε όμως είναι πολύ, πολύπλοκος και ε, οι προσδοκίες και προβλέψεις δεν είναι πολύ ενθαρρυντικές. Θα πρέπει να υπάρξουν και επιπλέον μέτρα. Ε, το βρετανικό παράδειγμα είναι ενδιαφέρον, γιατί ο συνδυασμός του ETS με, με την, και σύνδεση με το ε, με την τιμή του άνθρακα ήταν επιτυχή στον τελευταίο χρόνο. Γι' αυτό θέλω να τονίσω ότι η Total ήδη ε, εξετάζει την, την ανάδειξη μιας νέας τιμής στα 30 δολάρια ανατόνο. Με τις νέες τεχνολογίες χρειαζόμαστε και νέες ε, ναι, υποβολή ενδιαφέροντο. Όμω θα πρέπει αυτό να γίνεται κατά κλάδο για να έχουμε και τη συμπληρωματικότητα μεταξύ ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη βελτιστοποίηση των πόρων και, και την ισορροπία. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει σχεδιασμό σε πολλά επίπεδα και σε τοπικό επιφερειακό επίπεδο να έχουμε τη βελτιστοποίηση του ε, χαρτοφυλακίου αυτού μεταξύ των διαφόρων μορφών ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη για τη διαχείριση των επικρατιών και του πόρου ΑΠΕ. Πολιετής προγραμματισμός λοιπόν για τους διαγωνισμούς εξαρτάται κυρίως από την ε, διαδικασία, τη συχνότητα και τον αριθμό των διαγωνισμών αυτών στα κρατημέλη. Γι' αυτό και είναι κρίσιμη σημασία για την βιομηχανία και τους ε, παρόχους ε, να έχουν τουλάχιστον μια, έναν τριετή ορίζοντα, να γνωρίζουν δηλαδή τους διαγωνισμούς, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τους κανόνες κατανομής πόρων. Η εισαγωγή των ΑΠΕ στο σχεδιασμό της αγοράς και αν αυξήσουμε το μερίδιο των ΑΠΕ ε, στον ηλιακό μείγμα 50% το 2030 μαζί και με το 27% των ΑΠΕ όλα αυτά σημαίνουν ότι θα έχουμε ε, περισσότερες ημέρες με ποσοστά κοντά στο 100%. Αυτό απαιτεί μεγαλύτερη ευελιξία στον ευρωπαϊκό σχεδιασμό αγοράς ε, και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικά τα σήματα τιμών για να ενθαρρύνουμε έτσι την ε, ευελιξία. Θα ξεκινήσω από το φυσικό αέριο. Καλά κάνετε, Πρόεδρε, και τον αναφέρατε αρχικά, Πρόεδρε. Το φυσικό αέριο αφορά πολλούς ε, καταναλωτές και έχει πολλά στοιχεία για να μας φέρει πολύ καλές λύσεις. Ε, για την χρήση των ΑΠΕ, αλλά και συμπληρωματικά στη χρήση τους. Μετά, ε, διαχείριση από πλευρά ε, ζήτηση. Βασική προτεραιότητα, μετά έχουμε αποθήκευση, συσσωρευτέ, με καλύτερες ευκαιρίε και δυνατότητε. Διαχείριση προσφοράς. Πρέπει να έχουμε και διαλύπουσα προσφορά ενέργειας σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές ε, όπου ας πούμε έχουμε πολύ ήλιο, πολύ αέρα, ε, τα Σαββατοκύριακα και το καθεξής. Αυτό είναι ένα ε, ωφέλιμο εργαλείο για να εξισορροπήσουμε την προσφορά και ζήτηση. Εμεί στηρίζουμε την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναθεωρηθεί αυτό ο μηχανισμό. Ωστόσο, υπάρχουν δύο προποθέσει. Η σταδιακή εξάλληψη του dispatch θα πρέπει να γίνει προτεραιότητα απομείωση. Δεύτερον, επαρκή αποζημίωση για τι ε, ε που έχουν ε, περικοπεί για να προστατεύσουμε του καταναλωτέ. κατανάλωση. Στην Total σίγουρα είμαστε υπέρ ενός εφημιστικού πλαισίου που θα υποστηρίζει την αυτοκατανάλωση. Αυτό το επιχειρηματικό μοντέλο θα έχει όλο και αυξανόμενο αντίκτυπο και θέλουμε να ε, υπάρξει διασύνδεση στην Ευρώπη και να έχουμε κατάλληλες υπηρεσίες στο υλικό χρήστη και καταναλωτή. Τώρα επανέρχομαι στα, στις τέσσερις καταληκτικές μου παρατηρήσεις. Οι συνέπειες που θα έχουμε με <laughs> καλά, ο συνδυασμός των ε, διαφορετικών ενεργειακών πόρων θα περιορίσουν το κόστος ε, στην χοντρική. Γι' αυτό η Επιτροπή καλά κάνει και λέει στα κράτη-μέλη να εξαλείψουν τις ρυθμισμένες τιμές και θέλουν να συσσωρεύσουν διάφορες μορφές ε, και πηγές εσόδων. Δεύτερον, Μία βιομηχανική ε, στρατηγική που θα δώσει κίνητρα για τις τεχνολογίες χαμηλού άνθρακα. Ηλιακοί συλλέκτες. Τα κίνητρα λοιπόν ε, τα, και τα φαινόμενα του παρελθόντος με την κινέζικη κυριαρχία δεν μπορούν να επαναληφθούν πρέπει να έχουμε νέα μοντέλα. Γι' αυτό είναι πήγον η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαμορφώσει μια ε, βιομηχανική πολιτική από πλευρά ε, προσφορά. Ε, η καινοτομία και έρευνα και ανάπτυξη έχουν θετικά αποτελέσματα, ενθαρρύνουν την επιχειρηματικότητα και αγωνιστικότητα, ιδίω ό,τι αφορά την μεταποίηση κεντρικά και αποκεντρωμένα συστήματα, πολύ σημαντικά όλα αυτά, όμως ε, πρέπει να δούμε και το κόστος και την οικονομική αποδοτικότητα. Τέταρτον, ψηφιοποίηση και σύγκληση. Γιατί ο σχεδιασμός της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας πάει χέρι-χέρι με την ε, ε, ψηφιακή επανάσταση και πρέπει να ε, κινηθούμε από κοινού με ισχυρούς αλγορίθμους και τα μεγάλα δεδομένα. Αυτά είναι τα συμπεράσματά μου. Thank ευχαριστώ πολύ. Ήσασταν εξαιρετικός. Τελευταία ομιλήτρια, η κυρία Μόνικα Μοραβιέτσκα, μέλος του ε, Πολωνικού Συνδέσμου Ηλεκτρισμού, εκπροσωπεί τις ε, μεγαλύτερες εταιρείε ηλεκτρικής ενέργειας τη Πολωνία, αλλά και την ε, βιομηχανία ενέργεια. Η κυρία Μοραβιέτσκα εργάζεται 10 χρόνια στον κλάδο της ενέργειας και οι επαγγελματικέ τη δραστηριότητες συνδέονται άμεσα με, την, με τον Πολωνικό Σύνδεσμο Ηλεκτρικής Ενέργειας. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, αγαπητοί ευρωβουλευτέ δεν μπορώ παρά να αρχίσω με ένα σχόλιο λίγο εκτός θέματος, αν μου επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε. Είμαι γυναίκα από την Πολωνία και η Διεθνή ημέρα της Γυναίκας δεν έχει πολύ καιρό που πέρασε και αν το γνωρίζετε, η Πολωνία είναι η, η μόνη χώρα του ε, που κατάφερε να έχει ίσες αμοιβέ ε, ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες, σύμφωνα με την έκθεση που έχω στα χέρια μου. Είναι για μία φορά λοιπόν καλό να είσαι Πολωνή. Υπάρχει η έκθεση αυτή από την PwC ε, που σύμφωνα με αυτή η Πολωνία θα επιτύχει ισότητα στις αμοιβέ ανδρών και γυναικών ε, πολύ συντομότερα από τις υπόλοιπες. Σε 100 χρόνια. 100 χρόνια νωρίτερα από τις ε, υπόλοιπες. Υπάρχουν δύο εξαιρέσεις βέβαια σε αυτό. Ισπανία, το έτος όπου η Ισπανία θα έχει ίσες αμοιβές ανδρών και γυναικών, σύμφωνα με αυτήν την έκθεση, είναι το 2230 και το άλλο άκρο η Γερμανία, 2297 θα επιτευχθεί ισότητα αμοιβών ανδρών και γυναικών. Γι' αυτό λοιπόν ε, νομίζω πως πρώτα θα καταφέρουμε να έχουμε χώρες που εξαρτώνται αποκλειστικά από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ε, και μετά ίσες αμοιβές ανδρών και γυναικών. Αυτά προς το εκτός θέμα σχόλιο. Επιτρέψτε μου τώρα να συνεχίσω. Φυσικά, ο στόχος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για το 2030 είναι ένας ε, ε, δεσμευτικός στόχος σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχουν εθνικοί δεσμευτικοί στόχοι. Είναι καλό λοιπόν αυτό να το γνωρίζουμε προς το παρόν. Τώρα, ε, θα αναφέρω σύντομα τέσσερα κύρια προβλήματα που νομίζω πως έχουμε. Υπάρχουν κάποιες προβλέψεις για το πότε θα επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι και η πλατφόρμα χρηματοδότησης που λειτουργεί ως τιμωρία για όσους δεν επιτύχουν τους στόχους ε, συνδέεται και με τις ε, μας και με τη βιομάζα. Τώρα, γιατί νομίζω πως δεν θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικός ο χαρακτήρας ε, των, της επίτευξης του στόχου αυτού. Καταρχάς, ο χώρος της ενέργειας ε, δεν εξελίσσεται γραμμικά. Ιδιαίτερα όταν κοιτάξουμε τις ε, χώρες ξεχωριστά. Αν δούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύνολο, ίσως υπάρχει γραμμική εξέλιξη. Όμως ε, βλέπουμε ότι υπάρχουν μεγάλη, μεγάλα χρονικά διαστήματα στο σχεδιακό, σχεδιασμό. Γι' αυτό αυτή η γραμμική πορεία δεν θα έπρεπε να δημιουργεί παραθυράκια για να μπουν αυτοί οι υποχρεωτικοί, δεσμευτικοί στόχοι ενέργεια για την κάθε χώρα. Χρειάζεται ευελιξία. Είναι, πιστεύω, η λέξη κλειδί αυτή, διότι η ευελιξία θα δώσει την ευκαιρία στα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν τι δυνατότητέ του με τον πιο αποδοτικό και οικονομικό τρόπο. Και η γραμμική ε, εξέλιξη είναι ε, εντελώ αντίθετη σε αυτό. Μετά. Εθνική ο κανονισμό λέει πω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει αποκλειστικέ αρμοδιότητες. Δεν θα υπάρχει δυνατότητα ε, εξέταση ούτε από, το, από τα κράτη-μέλη ούτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί λοιπόν χρειαζόμαστε ένα τέτοιο μέσο. Πρώτον, το να στηρίζουμε τις ανανεώσιμες πέρα από τις ε, χώρες ε, που είναι δωρητές, ας πούμε, δεν δίνει ωφέλη στις χώρες αυτές. Κρύβονται πολλά πίσω από αυτό. Η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχει νόημα μόνο όπου το κόστος είναι χαμηλό και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χάσει δισεκατομμύρια ευρώ ε, επειδή ακριβώς δεν ακολούθησε αυτό το σκεπτικό. Στο μέλλον όμως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα πρέπει να εξαρτώνται από την αγορά, να βασίζονται στην αγορά. Τώρα μπορεί να μην μας αρέσει αυτό που ακούμε, μπορεί να προσπαθούμε να κάνουμε το αντίθετο, όμως πιστέψτε με θα γίνει. Θα βασίζονται αποκλειστικά και μόνο στην αγορά. Δεν θα χρειαζόμαστε ούτε χρηματοδοτική πλατφόρμα, ούτε επιχορηγήσεις. Μετά η διασυνοριακή συμμετοχή. Το να κάνει τα κράτη-μέλη να πληρώνουν για να αναπτυχθούν ανανεώσιμε και υποδομέ σε άλλα κράτη-μέλη νομίζω πω είναι λάθο οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πρέπει φυσικά να ε, αναπτύσσονται εκεί που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αλλά δεν νομίζω πως αυτό πρέπει να γίνει με επιχορηγήσεις και να προσπαθήσουμε να τεντώσουμε κάτι εκεί που δεν μπορούμε να το, να το χειριστούμε. Και πιστεύω ότι αυτή η υποχρεωτική, αυτό το υποχρεωτικό άνοιγμα των ε, επιχορηγήσεων ανάμεσα το 2021 και το 2025 νομίζω πως είναι υπερβολικό. Μετά, η βιομάζα. Η βιομάζα δεν θα πρέπει να, ε, δεν θα πρέπει να παραμελείται διότι είναι ένα πολύ σημαντικό μεταβατικό καύσιμο. Η βιομάζα είναι το καλύτερο μεταβατικό καύσιμο ε, για τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας που προσπαθούν να αποδεσμευτούν από τον άνθρακα. Και τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας με βιομάζα λειτουργούν συμπληρωματικά για τις ενδιάμεσες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ας μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή η βιομάζα παραμένει μεγαλύτερη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας στην Ευρώπη. Τέλος. Κάτι που ακούστηκε ήδη βέβαια είναι τα ε, πρότυπα επιδόσεων εκπομπών. Δεν θα σταθώ ιδιαίτερα σε αυτό, αλλά θα πω μόνο πως χρειάζονται φεδρικά ε, συστήματα και από θέματα ενέργειας, όχι μόνο τώρα, αλλά μέχρι τη στιγμή που αποκτήσουμε ε, επαρκή χωρητικότητα αποθήκευσης. Γι' αυτό λοιπόν το ETS νομίζω πως... το πρότυπο EPS δεν το χρειαζόμαστε. Υπάρχουν άλλοι μέθοδοι για να φτάσουμε σε αυτό το στόχο, διότι χρησιμοποιώντας το EPS ε, θα τεθεί σε κίνδυνο ο ενεργειακός εφοδιασμός σε ορισμένες χώρες. Δεν θα πω ποιες. Το περασμένο Σάββατο περίπου 20% της ε, του ενεργειακού μείγματος προερχόταν από την αιωλική ενέργεια. Στην ε, Πολωνία το ποσοστό αυτό έφτασε το 18%. 78 γιγαβατόρες. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά στην ε, Πολωνία έχουμε περισσότερη αιωλική ενέργεια από τη Δανία, που χρησιμοποιεί κατά κόρον αυτή τη μέθοδο παραγωγής ενέργειας. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μοραβιέκα. Τώρα περνάμε στον κύκλο των ερωτήσεων και των απαντήσεων, αρχίζοντα όπως και πριν με τους συζητητές και με πρώτο τον κύριο Κάριν, σχεδιασμό αγορά ενέργεια. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ρωτήσω μια απλή ερώτηση που αφορά τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργειας και τι επιχορηγήσει. Τι πρέπει να γίνει έτσι ώστε να αναπτυχθούν ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια χωρί να χρειαστούν επιχορήγηση. Πρέπει να είναι νέοι τύποι ανανεώσιμων αγορέ, χρειάζεται ε, διαφορετική νομοθεσία, είναι ρυθμιστικό το πρόβλημα, πρόβλημα τη αγορά. Πώ μπορούμε να αφήσουμε τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια να αναπτυχθούν, να εξελιχθούν χωρί να υπάρχει βοήθεια οικονομική. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Μπλάνκο Λόπες, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αρμόδιος ηγητής. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Δεν είναι τώρα το θέμα η ώρα να σχολιάσω διάφορα θέματα που θα προτείνω σε συζητήσει και που αποτελούν κομμάτι των ανησυχιών και όσων ανέφεραν ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να θέσουμε επιχειρήματα όσον αφορά τα σχέδια ισότητας γιατί ήμουν μέλος της Ισπανικής κυβέρνησης όταν, όταν πρώτη ενέκρινε νόμο περί ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών αλλά και ε, που επιτρέπει γάμο ε, μεταξύ ανθρώπων του ιδίου φίλου. Σας ευχαριστώ πολύ για τις εισηγήσεις σας. Ε, ε, βλέπουμε ότι η αγορά δεν δίνει σωστά μηνύματα όσον αφορά τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Ορίζει τις, αγορα... τις τιμές, αλλά δεν προσφέρει σαφή μηνύματα όσον αφορά τις επενδύσεις. Θεωρείτε πως είναι κατάλληλες οι προτάσεις ε, που παρουσιάστηκαν για να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Επίσης θέλω να σας ρωτήσω ποια είναι η θέση σας σε σχέση με την κατάργηση της προτεραιότητας της αποστολής και πρόσβασης σε ε, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ε, διανομής μάλλον και πρόσβαση σε ανανεώσιμες πηγές. γιατί θα πρέπει να απομακρυνθούμε από τις ρηπαίνουσες ε, πηγές προς τις καθαρές πηγές ενέργειας. Και όπως ήδη ακούσαμε σήμερα, η χειραφέτηση του πολίτη που προωθεί ο νέος κανονισμός είναι σπουδαίο νέο και θέλω να ρωτήσω ιδιαίτερα τον κύριο Δανόσο ε, ποιες είναι οι ευκαιρίες που προκύπτουν από τον συνδυασμό της αυτοκατανάλωσης και της ε, ε, μείωσης, μάλλον της ε, ε, εξέλιξης των συσσωρευτών, των στυλών συσσώρευσης και των εμποδίων που υπάρχουν για τη χρήση τους. Ο κύριος Τούρμες, ευχαριστώ. Πρέπει πρώτα να πω ότι ακόμα δεν έχω συνηθίσει το γεγονός ότι το ΤΑΛ τελικά είναι ο πιο μεγάλος Παραγωγό ηλιακή ενέργειας στην Ευρώπη, ο πιο μεγάλος παραγωγός μπαταριών στην Ευρώπη και μόλις αγόρασε και έναν ε, παραγωγό ε, πράσινη ενέργεια. Αλλά βρίσκω ότι αυτό είναι καταπληκτικό γιατί δείχνει ότι ο παλαιός κόσμος της ενέργειας κατάλαβε πως υπάρχει ένας νέος κόσμος της ενέργειας. Ε, τώρα, πώ χειρίζεσαι το Carbon Flow Price. Ε, ε, ε, έχουμε μια τεράστια, τεράστιο πρόβλημα στην αγορά. Γιατί και πώς θα μπορούσε αυτό να βοηθήσει. Και έπειτα τα μεγάλα εμπορικά κτίρια. Εκεί οι ηλιακοί, οι ισορρευτές και όλα μαζί θα μπορούσαν να συνδυαστούν θετικά. Ευχαριστώ για το καταπληκτικό μάθημα που κάνατε για την ισότητα των φίλων, κύριε μου. Όμως εσείς συνειδητοποιείτε ότι έχετε, ε, αντιφάσκετε στις δηλώσεις σας. Εσείς ζητάτε επιδοτήσεις για το νέο άνθρακα, παρά το γεγονός ότι πριν από 10 χρόνια το G20 είπε βασικά Ας καταργήσουμε τις επιδοτήσεις. Το 550 τι σημαίνει. Σημαίνει την παρεμπόδιση νέων επιδοτήσεων στην Πολωνία για τον νέο άνθρακα. Ζητάτε επιδοτήσεις για τον νέο άνθρακα και μετά λέτε ότι οι ανανεώσιμες δεν θα πρέπει να παίρνουν επιδοτήσεις. Αυτή είναι μια αντίφαση που δείχνει απλά πόσο ασυνεπή είναι η σκέψη σας. Και έπειτα μία πρόταση προς τον πολωνικό ε, τομέα ηλεκτρισμού. Όταν δείτε τις τιμές 49 ευρώ ανά μεγαβατόρα Ξέρω ότι η PG έχει προχωρήσει πολύ για ε, αιωλική ενέργεια στα ανοιχτά της θάλασσας. Εάν χρησιμοποιηθούν ευρωπαϊκά χρήματα για να μειωθεί το κόστος του περάσματος των καλωδίων, δεν θα ήταν αυτή μια από τις σπουδαιότερες ευκαιρίες για την Πολωνία και το πολωνικό τομέα ηλεκτρισμού να έχουν 3, 4, 500 ΜΒ σε εγκαταστάσεις αιωλικής ενέργειας στην ανοιχτή θάλασσα χιλιάδες θέσεις απασχόλησης. Δεν είναι αυτή η λύση για να ξεφύγετε από το, την πολύ δύσκολη κατάσταση που βρίσκεστε. Ευχαριστώ πολύ κύριος Ρόιλ. Ερώτηση. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να μου απαντήσετε, όποιος από τους τρεις θέλει, πώς ε, νομίζετε πως πρέπει να είναι οι στόχοι, αν χρειάζονται ε, υψηλότεροι στόχοι για τις ανανεώσιμες διαφορετικές προθεσμίες, χρονοδιαγράμματα. Θεωρείτε πως μέσω πρόθεσμα μπορούμε να αντέξουμε ε, με τις συμφιστάμενη συνθήκες στην Ευρώπη ή μπορούμε να είμαστε και πιο γρήγοροι στην ε, μετανοικιακή μετάβαση. Και μετά θα ήθελα, αν μου απαντήσετε αυτό το σκέλος, να μου πείτε και πώς φαντάζεστε ότι θα γίνει αυτό. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Γκροστέτ. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ σύντομα, κύριε Πρόεδρε. Η Επιτροπή στην αναθεώρηση τη οδηγία των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια προτείνει πραγματική τεχνολογική ουδετερότητα στις, ε, στην πρόσκληση που βλέπει ενδιαφέροντο. Όμω, ο σκοπός δεν είναι να παίρνουμε τον λιγότερο ε, δαπανηρό, αλλά να λαμβάνουμε υπόψη μια σειρά κριτηρίων, όπως είναι για παράδειγμα και η αποδοχή από την τοπική κοινωνία. Αυτό θα επέτρεπε να έχουμε μια πραγματική πολιτική βιομηχανικό τομέα. Εσείς θεωρείτε ότι αυτή η τεχνολογική ουδετερότητα ε, που είναι απαραίτητη πλέον ε, στις, στην πρόσκληση που πολύ ενδιαφέροντος μπορεί να έρθει ε, αντιμέτωπη και να παρεμποδίσει την ανάπτυξη αυτών των κλάδων της βιομηχανίας. Ευχαριστώ κύριε Λεπαντόφσκι. Προ την κυρία Μοραβέτσκα, βεβαίω δεν σα προκαλεί έκπληξη. Ευχαριστούμε για την προειδοποίησή σα. Έχει έρθει η ώρα οι άντρε να περασπιστούν την ισότητα μεταξύ των φίλων στην Πολωνία και είμαστε έτοιμοι. Αλλά σας ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας σε ό,τι αφορά την χρηματοδότηση των πόρων από τα κράτη-μέλη που δεν τα πηγαίνουν τόσο καλά. Δεν είναι μεθοδολογία του μαστιγίου και του καρότου, πρόκειται μόνο για το μαστίγιο. Σε αντίθεση λοιπόν με την έννοια της δημοσιονομικής ικανότητας για την Ευρωζώνη που δίνει ε, επιβραβεύσεις, αυτό είναι κάτι το διαφορετικό θα μπορούσαμε να επηρεάσουμε τα κράτη-μέλη να θεσπίσουν λιγότερο φιλόδοξους στόχους για να αποφύγουν τις οικονομικές κυρώσεις. Επομένω, θα υπήρχε έτσι ένα χάσμα φιλοδοξίας ε, σε κάποια κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριο Σκουλέτς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω τον τίτλο της σημερινής ε, ακρόασης και να ρωτήσω πού είναι οι Ευρωπαίοι πολίτες στους οποίους αναφέρουμε στον τίτλο. Το βασικό μήνυμα της Κομισιόν είναι ότι οι πολίτες βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της ενεργικής μετάβασης και της, πακέτου και της δέσμης μέτρων. Δεν άκουσα όμως τίποτα ε, σε ό,τι αφορά την συλλογική παραγωγή ενέργειας ε, ε, για τις απέπουν διαθέσιμες προς τους πολίτες, προτεραιότητες σύνδεσης στο δίκτυο, παραγωγή θερμότητας γιατί είναι σημαντικό τμήμα ε, του πακέτου αυτό, η θέρμανση και η ψήξη. Ε, το ίδιο ερώτημα προς όλους τους ομιλητές. Ευχαριστώ κυρία Νίμπλερ. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Η ερώτησή μου είναι πολύ συγκεκριμένη και απευθύνεται σε όλους σας, σε όποιον μπορεί να την απαντήσει, όποιος είναι κατάλληλος. Η οδηγία θα συμπεριλάβει και τη δασοκομεία. Για πρώτη φορά υπάρχουν κάποια κριτήρια βιωσιμότητα τα οποία προβλέπονται και για την ε, βιώσιμη διαχείριση των δασών. Αυτό δεν το καταλαβαίνω και αναρωτιέμαι αν είναι πραγματικά αναγκαίο. Διότι όλες οι αναλύσεις μας μέχρι τώρα και οι αναλύσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οδηγούν στο ίδιο συμπέρασμα ότι η δασοκομεία ε, δεν ε, αντιμετωπίζει προβλήματα, δεν υπάρχει κίνδυνος για τη βιωσιμότητα. Γι' αυτό λοιπόν αναρωτιέμαι γιατί εμείς τώρα ε, δημιουργούμε περισσότερο, περισσότερη γραφειοκρατία με τη συμπερίληψη και της ασοκομείας. Θα μπορούσε κάποιος από εσάς να μου απαντήσει. Αν υπάρχουν κάποιοι ε, σωστοί λόγοι, κάποια αιτιολογία. Σας ευχαριστώ πολύ. Κάλε. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, θα ήθελα... Μου άρεσε μάλλον που ακούσαμε όλα αυτά για την ισότητα των ε, φίλων στην Πολωνία. Κάποιος ξέχασε να τα πει όλα αυτά στον συνάδελφο κύριο Μίκη, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Είναι πολλά τα στήματα που πρέπει να εξετάσουμε, καθώς ε, και τα βιοκαύσιμα, σε παραγωγή κτλ. Πρέπει να τα εξετάσουμε και θα λάβουμε σίγουρα μια επικοδομητική στάση. Όμω δεν είναι σωστό αυτό που είπατε ότι μπορεί να έχουμε πετύχει τον ε, στόχο το 27% για τις ΑΠΕ. Πρώτον, γιατί ο κύριος Γιούγκερ ξεκαθάρισε ευθύ εξ αρχή ότι ήθελε η Ευρώπη να, είναι, ε, να έχει την ηγετική θέση στις ε, ανανεώσιμε και δεύτερον, πολλοί εδώ στο Κοινοβούλιο θεωρούν ότι το 27% είναι πολύ χαμηλό χάρη στην πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι σήμερα, χωρίς καμία απολύτως ε, προσπάθεια, φτάνουμε το 23% μάλλον. Οπότε το 27% δεν φτάνει. Προτείνεται ενδεχομένως ακόμα και να φτάσουμε στο 30%, αλλά αυτό είναι προσυζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κρασνοντέμσκι τώρα. Ο κύριος Τούρμες ήταν ιδιαίτερα αισιόδοξο σε ό,τι αφορά το μέλλον της Πολωνίας. με ένα τεράστιο όγκο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά ξεχνάτε πόσα χρόνια πήρε η ανοικοδόμηση στη Γερμανία, για παράδειγμα, ε, όπου μέχρι πρόσφατα χρησιμοποιούσαν σε λιμένες, άνθρακα κτλ. και μας είπαν ότι η τεχνολογική καινοτομία θα πάρει 25-30 χρόνια στη Γερμανία. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω την κυρία Μοραντιεύσκα ποια θα είναι η επίπτωση, ποιε θα είναι οι συνέπειε στην πολωνική αγορά ενέργειας που θα προκύπτουν από αυτά τα νέα πρότυπα εκπομπών που προτείνονται σε αυτή τη δέσμη. Ενδεχομένως η απάντηση να είναι αυτή που έδωσε συνάδελφος προηγουμένως, ότι κάθε χώρα θα πρέπει να ε, αναλάβει τη δική της επικράτη και να λύσει τα δικά της προβλήματα. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ε, δεν βλέπω κάποιος άλλος να ζητάει τον λόγο. Να προσθέσω εγώ δύο πράγματα. Πρώτον, θεωρείτε ότι υπάρχει κάποια προοπτική και πότε νομίζετε ότι θα φτάσουμε στο σημείο να μην χρειαζόμαστε επιδοτήσεις ε, και ενισχύσεις ε, για ορισμένες ε, μορφές ενέργειας και για τις ανανεώσιμες. Εξετάζοντα την Ενεργειακή Ένωση και Αγορά Ενέργεια το 2013, είχαμε μιλήσει για τον οριζοντα ορίζοντα 2020-2022. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό ισχύει πια. Βέβαια αυτό δεν αφορά μόνο τι ανανεώσιμε, αλλά όλες τις πηγές ενέργειας. Δεύτερον, λίγο προκλητικά, μήπως υπάρχει περίπτωση οι αγορές ικανότητας κάπως να δώσουν κίνητρα στην ε, ανάπτυξη των ΑΠΕ, γιατί κάποιες φορές ε, ακούω κάτι τέτοια. Και αν ναι, υπό ποιες περιποθέσεις και πώς γίνεται να γίνει κάτι τέτοιο. Και ίσως η κυρία Μοραβέτσικα μπορεί να το απαντήσει, γιατί εσείς δεν το θίξατε. Δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις από ό,τι βλέπω, οπότε να σας δώσουμε το λόγο να απαντήσετε. Εσείς θα καθορίσετε με ποια σειρά θα απαντήσετε. Ξεκινήστε. Ωραία. Total. Yes. I will try to answer to your question regarding... Θα προσπαθήσω να απαντήσω στην ερώτησή σας σε σχέση με τις επιδοτήσεις. Είναι σίγουρα το δυσκολότερο και όλοι ονειρευόμαστε το δισκοπότηρο, το ιερό δυσκοπότηρο. Στο παρελθόν ήταν εύκολο διότι το περιθωριακό ηλεκτρόνιο από το περιθωριακό παραγωγικό εργοστάσιο ε, ε, θέσπιζε την τιμή. Τώρα τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Τώρα χρειάζονται επιδοτήσεις για όλες τις ενέργειες στην ε, παραγωγή ηλεκτρισμού. Αν είναι μόνο ένα σύστημα ενέργειας, το χρειάζεσαι για την πυρνική ενέργεια. Τώρα τρεις φορές περισσότερο κοστίζει από την ηλιακή ενέργεια. Ε, τέλος πάντων δυόμιση φορές περισσότερο κοστίζει. Οπότε Πρέπει λοιπόν να αναδιατυπώσουμε τη θεωρία. Τη θεωρία δεν την έχουμε φτιάξει ακόμα και πρέπει μετά να κάνουμε προσωμιώσεις, κοιτώντα ίσως πέντε χρόνια πριν ποια ήταν η ζήτηση, ποια θα ήταν η κατάσταση ε, για το 2030 και να δούμε ένα δευτερόλεπτο ή ένα λεπτό και να προσωμιώσουμε στα, για τα επόμενα πέντε χρόνια με τον αντίστοιχο καιρό για να δούμε αν θα είχαμε 100% ηλεκτρισμό στη σωστή στιγμή και στη σωστή θέση. Μπαίνουμε σε ένα πολύ περίπλοκο κόσμο, δεν έχω τη λύση. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι στο μέλλον η ηλιακή θα είναι, τα φωτοβολταϊκά θα είναι φθηνότερη. Αν δούμε τη Δανία ή τη Γερμανία και την Πορτογαλία ή την Νότια Ισπανία, είναι ήδη 1 ευρώ που είναι αντίστοιχο με το 30 ευρώ. Μπορούμε να το σκεφτούμε αυτό για τα επόμενα 30 χρόνια. Δηλαδή σταθερή τιμή στα 30. Όχι. Πολύ περίπλοκο το σύστημα και δεν έχω μια απάντηση γιατί θα πρέπει να φτιάξουμε μια κάποια θεωρία για να μπορέσουμε όλα αυτά να τα αντιμετωπίσουμε. Και αυτό ανέφερα και στο παρελθόν, και στην αρχή μάλλον συζητησή μου, όπως και στις μπαταρίες. Πρέπει να δούμε διαφορετικές ροές εσόδων, γιατί αν έχουμε μόνο για τις ε, συσσωρευτές ενέργεια, η χωρητικότητα δεν είναι οικονομικό να μπουν οι συσσωρευτές στο σύστημα τώρα. Εάν συνδυάσουμε την αξία της ενέργειας που αποθηκεύεται ή τη χωρητικότητα των βοηθητικών υπηρεσιών από το πλέγμα, για παράδειγμα, τότε φτάνουμε στη σημερινή οικονομία. Αυτό για να απαντήσω στην ε, ερωτήσεις σας. Αυτή είναι και η πρώτη σας ερώτηση σε σχέση με τον πυρηνική, τον άνθρακα. Πρέπει να δουλέψουμε, πιστεύω, πολύ σκληρά. Απλή απάντηση, ναι, χρειαζόμαστε επιδοτήσεις στο μέλλον. Αλλά όλα τα ίδια ενέργειες στο πλέγμα. Αυτό ξέρω ότι είναι προκλητικό απάντηση, αλλά πρέπει να το δούμε με διαφορετικό τρόπο και να μην σκεφτούμε τις επιδοτήσεις. Είναι ε, ένα νέο σχεδιασμό του συστήματο αγορά. και η λέξη επιδότηση δεν ταιριάζει εδώ. Which has carbon... Carbon Flow Price είπατε. Ε, νομίζω πως είναι μία λύση είναι μια μερική λύση. Η αγορά των εκπομπών, της εμπορίας εκπομπών δεν θα δίνει στη σωστή στιγμή το σωστό μήνυμα, το σωστό σήμα. Θα πάρει χρόνια μέχρι ότου έχουμε το σωστό σήμα. Σήμερα η αγορά είναι στα πέντε και μπορούμε να προβλέψουμε από την απόφαση του, τρι, του τριμερούς. Όλοι το γνωρίζουμε αυτό, οπότε δεν αρκεί. Κάτι πρέπει να προσθεθεί. Carbon Flow Price στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει αποδείξει ότι είναι επιτυχές. Θα πρέπει να, είναι μια λύση που θα πρέπει να τη σκεφτούν κάποια κράτη-μέλη. Μιλήσατε για τα μεγάλα εμπορικά κτίρια, ναι, οπωσδήποτε. Αλλά θα είχα να προσθέσω το εξή. Αυτό που έρχεται τώρα είναι ότι όλοι, εγώ και εσείς, ως τελική χρήστης καταναλωτές μπορώ να είμαι καταναλωτής και μπορώ να έχω στην ε, ε, σκεπή μου ε, φωτοβολταϊκά και να έχω και ένα ηλεκτρικό όχημα και να βελτιστοποιήσω το σύστημά μου, να ελαχιστοποιήσω το κόστος μου. Θα είναι πολύ περίπλοκο. Μετά θα υπάρξουν νομοδοποιητές που θα έρχονται και θα δίνουν τις λύσεις. Και μετά αυτοί οι άνθρωποι θα αναμεγνύονται μάλλον με την ασφαλιστική εταιρεία, την Telecom, την Google και θα προσπαθήσουν λοιπόν να ομοδοποιήσουν τις υπηρεσίες ώστε να μεγιστοποιήσουν τα έσοδα από το B στον C, δηλαδή και από τον καταναλωτή αλλά και από τα μεγάλα εμπορικά κτίρια. Σίγουρα λοιπόν είναι ευκολότερο σήμερα οι λύσεις που συνδυάζουν τα φωτοβολταϊκά με τους συσσωρευτές, με τη διαχείριση ζήτησης και προσφοράς, με καλούς αλγορίθμους και σίγουρα για τα εμπορικά κτίρια. Ήδη γίνεται και θα αναπτυχθεί ε, ακόμη περισσότερο, σίγουρα. Και αρκετές εταιρείες ε, ασχολούνται με αυτό το τομέα. Είναι θετικό. ουδετερότητα στις ε, τεχνολογικούς ε, διαγωνισμούς, ε, ναι βεβαίως. Είμαστε κατά αυτής της τεχνολογικής ουδετερότητας, διότι δεν μπορεί να υπάρχει η ανανεώσιμη ενέργεια είναι μια εδαφική ενέργεια. Σε αυτή την περιφέρεια δεν έχει απαραίτητο ε, αέρα ή μπορεί να έχει και αεολική και, και ηλιακή. Και, και αυτό είναι καλό να τα συνδυάσει σε περιφερειακό ή σε κρατικό επίπεδο. Είναι πολύ καλύτερο λοιπόν το κράτος να μπορεί να διαχειρίζεται την επικράτειά του, το σχεδιασμό του και θα δώσει και στις διάφορους ε, ε, κλάδους τη δυνατότητα να ανταγωνιστούν παγκοσμίω. Γιατί η αιωλική ενέργεια πρέπει να ανταγωνιστεί και με την Κίνα. Τα ηλιακά, η ηλιακή ενέργεια είναι ήδη δύσκολο, υπάρχει ήδη μεγάλος ανταγωνισμός. Πρέπει να μπορούμε να είμαστε σε θέση και ελπίζω πως θα ε, ε καταπολεμηθεί αυτή η πρόταση. Δασοκομεία. Δεν μιλήσαμε για τα βιοκαύσιμα και αυτό μου δίνει μια λαβή. Ελπίζω, Πρόεδρε, πως θα με καλέσετε για να μιλήσουμε και για τα βιοκαύσιμα, τη δασοκομεία, όλα όσα συνδέονται με τη γεωργία και τη βιομάζα. Διότι πραγματικά εμείς στην Total πιστεύουμε πως μπορούν να γίνουν πολλές βελτιώσεις στην πρόταση της Κομισιόν για τα θέματα βιομάζας. Δεν θα τα συζητήσω σήμερα γιατί περισσότερο σήμερα είχαμε να μιλήσουμε για τον ηλεκτρισμό και το σχεδιασμό ε, και ελπίζω πως θα με καλέσετε όταν θα συζητήσετε και τα βιοκαύσιμα. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σαπερό, που είστε ε, αντιπρόεδρος της ΤΟΤΕΛ. Ο κύριος Δανόσο από τον ε, Ισπανικό Σύνδεσμο Φωτοβολταϊκών. Ευχαριστώ. Συμμερίζομαι πολλά από αυτά που είπε ο κύριος ε, Σαπέρο. Και ε, Πρώτα η χαρακτηριστική ερώτηση. Εγώ πάνω από 30 χρόνια είμαι στον κόσμο των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια και πάντα αυτή την ερώτηση ακούω. Πότε θα είναι ανταγωνιστικέ οι ανανεώσιμε, πότε δεν θα χρειάζονται πια επιδοτήσει. Τώρα που δεν τι χρειαζόμαστε, το πρόβλημα είναι ότι μα ε, ε, κρατάνε εκεί γιατί φοβούνται την ανταγωνιστικότητά μα και την αυτο, αυτοκατανάλυση. Οι ανανεώσιμε είναι ανταγωνιστικέ, αλλά πρέπει να ορίσουμε τι θα πει ανταγωνιστικότητα. Για παράδειγμα, μέσα σε ένα μήνα στη χώρα μας, στη χώρα μου, την Ισπανία, θα γίνει ένας πληστηριασμός. Πληστηριασμός για ε, την ανανεώσιμη ενέργεια. Αν δεν είχε τόσο χάλια σχεδιαστεί αυτή ο πληστηριασμός, μέσα σε ένα μήνα θα βλέπαμε τιμές ανά τώρα κάτω από τα 20 ευρώ για ένα μεγαβατόρα. Αν σκεφτούμε ότι 45 κόστιζε η μεγαβατόρα τα τελευταία χρόνια στην Ισπανία, μπορούμε να δεχτούμε πω ήδη αυτό σημαίνει ότι είμαστε ανταγωνιστικοί. Είμαστε ανταγωνιστικοί με βάση τι συνθήκε αγορά που επικρατούν αυτή τη στιγμή. Και όπω είπα, δεν είναι συνθήκε αγορα που επικρατούν αυτή τη στιγμή. Και οπω είπα, δεν είναι συνθηκε αγορα ιδανικε για τι ανανεώσιμε, για τα χαρακτηριστικά του. Αυτό είναι ένα από τα μεγάλα μειονεκτήματα αυτή τη πρώτη οδηγία, ότι δεν ρισκάρει βλέπουμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε προς ένα στόχο μέχρι το 2050 όπου αν δεν το πιστέψουμε, η οικονομία μας, ε, μάλλον ότι που πρέπει μάλλον η οικονομία μας να, να μην χρησιμοποιεί πλέον άνθρακα. Πρέπει να χαράξουμε έναν δρόμο, μια απορία και εδώ ε, συνδέομαι με το θέμα των στόχων. Πρέπει να φτιάξουμε λοιπόν μια ατζέντα που να δίνει ένα μήνυμα ότι πραγματικά θέλουμε να φτάσουμε στο 100% το 2050. Και αν το λέμε εδώ σε αυτό το κοινοβούλιο να λέγεται ότι φτάσαμε στο 27% τότε υποθέτουμε πως Στη συνέχεια αφήνουμε ε, τα καθήκοντά μας για τα επόμενα 20 χρόνια. Είναι λίγο πιστευτό ότι στα επόμενα 20 χρόνια θα κάνουμε το υπόλοιπο 73%. Χρειάζεται να θέσουμε ρεαλιστικούς στόχους ώστε να δώσουμε και τα κατάλληλα μηνύματα. Τουλάχιστον να φτάσουμε ένα 35%, ένα 40% και σιγά σιγά να προχωρούμε σε αυτό το δρόμο. Επιπλέον, αυτός ο στόχος του 27% είναι business as usual. Δηλαδή, δηλαδή το φτάνουμε χωρίς να κάνουμε τίποτα με αυτό το βαθμό ανταγωνιστικότητας. Είναι πολύ δύσκολο να σκεφτεί κανείς ε, ότι θα φτιάξει κάποια εγκατάσταση και να επενδύσει σε άλλο είδος ενέργειας εκτός από τις ανανεώσιμες. Όμως επιπλέον αυτός ο στόχος του 27% υπολογίστηκε σε απόλυτους όρους και με βάση έναν ε, στόχο απόδοσης της Ευρωπαϊκής Ένωση για 27%. Όμως αυτός ο στόχος έχει ήδη αυξηθεί στο 30% και θα αυξηθεί και περισσότερο. Δουλεύουμε με βάση χαμηλότερο αρχή. Θα ήταν πιο φυσικό να έχουμε ήδη ξεπεράσει το 30%. Και αυτό πρέπει να γίνει για να δώσουμε ένα σημάδι αξιοπιστία στον υπόλοιπο κόσμο. Ότι δηλαδή η Ευρώπη δεσμεύεται για την επίτευξη συγκεκριμένων περιβαλλοντικών στόχων και θα φτάσει τουλάχιστον στο 35% και να είναι δεσμευτική αυτή η στόχη. Γιατί? Γιατί είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι υπάρχουν κάποιες χώρες που λένε όχι, όχι, εγώ δεν θέλω να μου επιβάλλουν όρους θα το πετύχω το στόχο εγώ, αλλά χωρί όρου. Δηλαδή, τι κάνουμε στην ουσία, ανοίγουμε και ένα παραθυράκι για να μην τηρήσουμε αυτό το στόχο. Όλες οι χώρες ε, δεσμευτήκαμε ότι θα ε, θέσουμε στόχους που απότερο στόχος του θα είναι η επίτευξη του συνολικού στόχου για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, τεχνολογική εξέλιξη. Είναι προφανές ότι αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι έργα τα οποία είναι πιο ανταγωνιστικά, πιο σύμφωνα με την αγορά που έχουμε τώρα και που θα έχουμε. Αν όμως ταυτόχρονα θέλουμε να στείλουμε μήνυμα στο βιομηχανικό κόσμο, στον κόσμο της τεχνολογίας, ώστε η Ευρώπη ακριβώς να ακολουθήσει αυτό το δρόμο, αυτό θα είναι πλεονέκτημα ανταγωνιστικό, όχι μόνο για την καθαρή ενέργεια, αλλά γιατί έτσι χρειάζονται τεχνολογικές εξελίξεις. Να στείλουμε μήνυμα στην αγορά νέα αγορά σταθερή σε αυτές τις τεχνολογίες και αυτό ευνοεί και τις ιδιωτικές επενδύσεις και βοηθά στις ε, επενδύσεις στην τεχνολογία. Στον τομέα των φωτοβολταϊκών σχολιάστηκε πριν ε, το θέμα των συσσωρευτών, των φωτοβολταϊκών. Το, ε, ένα πάνελ φωτοβολταϊκό δεν σημαίνει παρά 30-35% του συνολικού κόστος του project. Δηλαδή υπάρχουν άλλα στοιχεία όπου υπάρχει προστεθέμενη αξία και όπου η ευρωπαϊκή βιομηχανία μπορεί να ειδικευτεί. Σχεδιασμός, ε, μετατροπής, ε, δομές, ε, όπου μπορεί να υπάρξει δηλαδή περισσότερη προστεθέμενη αξία για την Ευρώπη και όπου μπορούμε εμεί να παίξουμε σημαντικό ρόλο στον τεχνολογικό κόσμο των φωτοβολταϊκών, χωρίς να είναι μόνο τα πάνελ τα οποία είναι όλα ένα και μικρότερα και με μεγαλύτερη ακρίβεια όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα και την περιορισμό του κόστους και των περιθωρίων. Κόστος που από ό,τι προβλέπετε τα επόμενα χρόνια θα μειωθεί ε, κατά 20-25%. Και δεν θέλω να τελειώσω χωρίς να αναφερθώ στις ε, ε, κοινωνικές ε, συλλογικότητες στους συλλόγους των φωτοβολταϊκών. Για μας αυτό είναι απαραίτητο. Είναι ο τρόπος με τον οποίο ο κόσμος μπορεί να έχει πρόσβαση στα ωφέλη της κατανάλωσης των ενέργειας από τα φωτοβολταϊκά. Είναι τρελό ότι αυτή τη στιγμή απαγορεύει η ισχύουσα νομοθεσία αυτού του είδους την αυτοκατανάλωση. Αυτή η απαγόρευση δεν γίνεται να υπάρχει. Δεν μπορεί να απαγορεύεται στον καταναλωτή, στον πολίτη να συγκεντρωθεί σε ένα σύνδεσμο, μια ένωση για να μπορεί να ε, εκμεταλλεύεται την ίδια κοινή αιωλική ή φωτοβολταϊκή εγκατάσταση που θα τους δίνει την ενέργεια που θα καταναλώνει η ίδια. Αυτό είναι σαφές, είναι ξεκάθαρο χειραφέτηση του πολίτη, αυτό το ωραίο σύνθημα, η ε, χειραφέτηση του καταναλωτή σημαίνει πραγματικά ότι θα πρέπει μπορεί να το κάνει. Και η συλλογική κατανάλωση είναι μια αποτελεσματική μορφή μετατροπ... Ε, πρακτικής μετατροπής αυτού του συνθήματος σε πραγματικότητα. Ευχαριστώ. Κυρία Μοραβιέσκα. Από τον, ε, την Πολωνική Ένωση Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ευχαριστώ πολύ. Επιτρέψτε μου να προσθέσω και εγώ δύο λόγια για το γιατί οι ανανεώσιμε δεν χρειάζονται επιχορήγηση. Συμφωνώ απόλυτα καταρχά με αυτά που είπε ο κ. Σαπερών. Πρέπει να δούμε τα πράγματα αλλιώ. Ε, δεν μπορούμε καταρχά να ε, δούμε το θέμα τη τιμή ε, συνολικά, αλλά πρέπει να δούμε το κόστο που βασισμένο σε πολλού επιμέρου τομεί και να δούμε το κόστο σε όλο τον κύκλο ζωή της ενέργειας. Και συμφωνώ εδώ ότι σε ορισμένες αγορές η ηλιακή ενέργεια θα είναι η πιο φτηνή πηγή ενέργειας. Γιατί λοιπόν να χρειάζεται επιχορήγηση. Χρειάζεται αυτή τη στιγμή επιχορήγηση διότι έτσι όπως είναι η αγορά υπάρχουν στρεβλώσεις. Αυτό είναι. Μόνο αυτό. Πρέπει να διορθώσουμε το πρόβλημα. και είναι πρόβλημα τώρα, όμως είμαι σίγουρη πως έχουμε τη δυνατότητα να το διορθώσουμε στο μέλλον. Είμαι σίγουρη λοιπόν, και το ξαναλέω αυτό, ότι κάποια στιγμή στο μέλλον ε, θα χρησιμοποιούμε αποκλειστικά και μόνο ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μόλις έχουμε την ε, ε, κατάλληλη τεχνολογία, μόλις πέσει το κόστος, μόλις αποκτήσουμε επαρκείς εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας. Δεν ξέρω πότε θα γίνει αυτό, θα γίνει όμως σίγουρα. Τώρα, για να απαντήσω στην ερώτηση του κυρίου Τούρμες για αυτές τις ασυνέπειες. Δεν ζητώ αυτή τη στιγμή επιχορηγήσεις για τον νέο άνθρακα. Το, ε, το EPS όπως είναι τώρα ε, εξαιρεί και τον άνθρακα που ήδη υπάρχει και τον νέο άνθρακα. Μπορώ όμως να σας απαντήσω στην ερώτηση του τι σημαίνει αυτό για την Πολωνία. Blackout. Αυτό θα σημαίνει. Θα χάσουμε στην ουσία το μεγαλύτερο κομμάτι της χωρητικότητάς μας, τις 55 μεγαβατόρες. Γίγαβατόρες. Και αν νομίζετε πως μέσα στα επόμενα χρόνια μπορούμε να αντικαταστήσουμε ε, ούτε έστω τις μισές από αυτές, 25 γίγαβατόρες, τότε ε, πλανόμαστε. Πλάνη νυχτεράνε. Τι μπορούμε να κάνουμε με το χειμερινό πακέτο, αν προσέξατε, υπήρχε και μια τελική έκθεση ε, που αφορούσε την έρευνα για την αγορά χωρητικότητας ηλεκτροπαραγωγής. Και ακούσαμε επανελειμμένα ότι η αγορά αυτή πρέπει να είναι ουδέτερη ως προς την τεχνολογία. Και αυτό είναι ως απάντηση σε αυτό που με ρωτήσατε, δηλαδή κατά πόσο θα υποστηρίξουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας χωρές. Θα τις υποστηρίξουν παρέχοντας δηλαδή την εφεδρική ικανότητα αποθήκευσης, είτε αυτό είναι άνθρακας, είτε αυτό είναι φυσικό αέριο, ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν, τις καιρικέ στο έδαφος κάθε ε, χώρας, ε, θα διαφέρει και η ικανότητα αποθήκευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Πρέπει να αποκτήσουμε μεγαλύτερε καταστάσει αποθήκευση, διαφορετικά δεν μπορούμε να έχουμε ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Δεν υπάρχει λοιπόν κάποια συνέπεια εδώ, ούτε επίση ε, ζητούμε να μην επιχορηγούνται οι ανανεώσιμε. Εμεί απλά είπαμε ότι δεν θα χρειαστεί να επιχορηγούνται γιατί θα είναι πιο φθηνέ. Και ε, κάτι άλλο που ίσως σας εκπλήξει, Εργάζομαι λοιπόν για τον Πολωνικό Σύνδεσμο Ηλεκτρικής Ενέργειας ε, ε, και για την PGE και με γνωρίζουν στην PGE ως υπέρμαχο των ε, offshore έργων, των υπεράκτιων έργων. Θεωρώ λοιπόν πως είναι ένα πολύ καλό έργο, πρέπει να το στηρίξουμε και ελπίζω να στεφθεί με επιτυχία. Δεν είναι βέβαια δική μας αποκλειστικά η απόφαση, αλλά υπάρχουν ευρωπαϊκά κονδύλια για τις υποδομές, οι οποίες αποτελούν ένα μεγάλο κομμάτι του κόστους. Συμφωνώ λοιπόν σε αυτό απόλυτα και χαίρομαι που συμφωνούμε σε κάτι. Τι άλλο, τι άλλο, ναι. Το καρότο και το μαστίγιο, η χρηματοδοτική πλατφόρμα, σίγουρα είναι μαστίγιο. Και αναρωτιέμαι γιατί το μαστίγιο βρίσκεται ακριβώς στους στόχους των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και όχι στους στόχους της ενεργειακής απόδοσης. Θα έπρεπε να υπάρχουν δεσμευτικοί ευρωπαϊκοί στόχοι και αναρωτιέμαι λοιπόν ποια είναι, ποιος είναι ο λόγος της ύπαρξής του στις ανανεώσιμες. Μετά, τα κράτη-μέλη γνωρίζουν πως αν δεν ακολουθήσουν την σχεδιασμένη πορεία θα υπάρξουν κυρώσεις. Και αυτό δεν είναι φιλοδοξία, το να κάνεις ό,τι χρειάζεται για να μην υπάρχουν συνέπειες. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή αρκετά σαφείς διατάξεις στον κανονισμό για τη διακυβέρνηση και χρειάζεται περισσότερη σαφήνεια. Χρειάζεται ε, σίγουρα να διορθωθεί αυτή η ασάφεια. Αλλά σίγουρα βρίσκω πως υπάρχουν λήψεις φιλοδοξίες. Δεν ξέρω αν ξέχασα κάτι. Νομίζω όχι. Νομίζω τα κάλυψα όλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε όλοι. Ε, νομίζω πως είδαμε πως έχει γίνει εξαιρετική δουλειά. Υπάρχουν πολλές νομοθετικές προτάσεις, η οδηγία για τις ανανεώσιμες έχουμε 7 εισηγητές. Και ακριβώς επειδή ενώσαμε στην έκθεση αυτή δύο διαφορετικές οδηγίες και έχουμε πολύ στενή συνεργασία, καταφέραμε ο συντονισμός να είναι πάρα πολύ καλός. Είναι η μεγαλύτερη δέσμη μέτρων στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο στον χώρο της ενέργειας, η μεγαλύτερη σε όλους τους τομείς. Πολύ σημαντική λοιπόν πρόταση ενώπιών μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που τη στηρίζετε με το έργο σας και ένα θερμό χειροκρότημα για τους προσκεκλημένους μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ε, dear friends. Αγαπητοί φίλοι, αύριο μπορούμε να συνεχίσουμε. Αύριο πρωί θα γίνει μια συζήτηση για την έκθεση Τούρμε σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και την έκθεση Γκέρεκε αναθεώρηση της οδηγίας ενεργειακής απόδοσης. Είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος. Ηλεκτρισμός, καθαρή ενέργεια, χειμερινό πακέτο δέσμη μέτρων, πείτε το πώς θέλετε. Σας ευχαριστώ πολύ.